Ε, members, ε, Αξιότιμα μέλη, έχουμε ήδη χάσει 8 λεπτά από το χρόνο ε, που θα είναι εδώ μαζί μας η Επίτροπος Τάισεν. Θα σας δώσω ευθύς αμέσως το λόγο κυρία Τάισεν και στη συνέχεια θα μιλήσει ο εισηγητής και οι σκιώδεις εισηγητές για δύο λεπτά ο καθένας. Έχετε το λόγο κυρία Τάισον. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη, είναι χαρά μου που βρίσκομαι εδώ σήμερα όπως πάντα στην Επιτροπή Απασχόλησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορώ να σας υποβάλω την πρότασή μου για την αναθεώρηση των κανόνων σχετικά με το συντονισμό για τα ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης. Ξέρετε ότι ο φάκελος αυτός θεωρείται νομοθετική προτεραιότητα στην κοινή δήλωση των τριών θεσμικών οργάνων και θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τον εισηγητή, τον κύριο Μπάλας, του εύχομαι και σε αυτόν και στους ε, σκιώδεις εισηγητές κάθε επιτυχία έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε γρήγορα πάνω σε αυτό το ζήτημα. Όταν ρωτάει κανείς τους Ευρωπαίους ποιο είναι το, το δικαίωμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο το οποίο ε, τους ε, ενδιαφέρει περισσότερο είναι η ελεύθερη κυκλοφορία, η απάντηση. Δεν θα ήταν εφικτή όμως αυτή η κινητικότητα χωρίς ε, ε, κανόνε σχετικά με τα συστήματα κοινωνική ασφάλισης και τον συντονισμό του. Αυτό είναι που εγγυάται ότι δεν θα χάσουν τα κοινωνικά του δικαιώματα, την κοινωνική του προστασία οι πολίτε όταν πάνε από μια χώρα στην άλλη. Βεβαίω τα κράτη-μέλη έχουν την απόλυτη ευθύνη και για το σχεδιασμό αλλά και για την οργάνωση των συστημάτων κοινωνική ασφάλιση. Αυτό άλλωστε προβλέπει και η συνθήκη. Οι διατάξει του κανονισμού αυτού καθορίζουν απλώς ε, σε ποιο σύστημα ανήκει ο κάθε ε, πολίτης ο οποίος μετακινείται. Ο χρυσός κανόνας είναι ότι πρέπει πάντα να καλύπτονται από ένα σύστημα και μόνο οι πολίτες. Είναι ε, η αρχή του ενιαίου συστήματος κάλυψης. Και εκεί συνήθως είναι που μπορούν να ζητήσουν και, τα, και τις τα όποια επιδόματα. Είναι ένας κανόνας που υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και απλώς την επικαιροποιούμε. Τώρα, γιατί χρειάζεται νέα επικαιροποίηση αυτή τη στιγμή. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, μια σειρά από οικονομικές ε, και κοινωνικές εξελίξεις. Οι εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, αυτοί που έχουν αναλάβει να εφαρμόσουν και να ερμηνεύσουν τους κανόνες αυτούς καθημερινά ε, συνήλθαν στα πλαίσια μιας διοικητικής επιτροπής. Εμείς προτείνουμε λοιπόν και προτείνουμε κάποιες τροποποιήσεις σε μια σειρά από τομείς. Τα επιδόματα ανεργίας καταρχήν. Να μπορεί κάποιος να μεταφέρει τα επιδόματα ανεργίας του, το επίδομα ανεργίας του σε μια άλλη χώρα για έξι μήνες αντί για τρει που ισχύει τώρα. Γιατί το προτείνουμε αυτό. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ένα εκατομμύριο άτομα που ψάχνουν θέσεις απασχόλησης σε άλλη χώρα από τη δική τους. Σε κάποιες χώρες έχουμε ψηλά ποσοστά ανεργίας, σε κάποιες όλες, άλλες έχουμε σχεδόν πλήρη απασχόληση και υπάρχουν και ελλείψεις μάλιστα, είναι λογικό να, είναι, να υπάρχει κινητικότητα και είναι επιθυμητό να υπάρχει κινητικότητα των εργαζομένων. Αλλά πρέπει να είναι, μπορούν να μετακινηθούν με βάση ίσους κανόνες, δίκαιους κανόνες για όλους και που να μην επιτρέπουν σε κάποιον να επιλέγει ό,τι θέλει. Όταν κάποιος λοιπόν δικαιούται ένα επίδομα ανεργίας στην χώρα όπου εργάστηκε για τελευταία φορά, θα πρέπει αυτό το επίδομα να μπορεί να το μεταφέρει για τουλάχιστον έξι μήνες και όχι τρεις όπως ισχύει σήμερα εφόσον θεωρεί κάποιο ότι έχει περισσότερε πιθανότητε να βρει μια θέση απασχόληση σε μια άλλη χώρα. Αυτό δεν είναι ότι ο καθένας επιλέγει ό,τι θέλει. Έχει συνεισφέρει ο άνθρωπος αυτό σε μια συγκεκριμένη χώρα με τις εισφορέ του και από εκεί λαμβάνει το επίδομα. Και βεβαίω υπάρχουν και προϋποθέσεις. Πρέπει το άτομο αυτό να έχει μείνει άνεργο ε, παρά τη θέλησή του και βεβαίω ε, το υπεύθυνο κράτο μέλος είναι αυτό που θα ελέγχει ε, ότι αυτά ισχύουν. Πρέπει εντό πολύ συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος να εγγραφεί στο νέο κράτος μέλος ε, ο εργαζόμενος ή ο πολίτης και θα πρέπει να υπάρχει μια αναφορά από το νέο κράτος μέλος προς το παλαιό για τι προσπάθειες του πολίτη αυτού στα πλαίσια της αναζήτησης εργασίας. Τώρα υπάρχουν και οι, άνθρωποι που ε, ζουν κοντά στα σύνορα, ε, ζουν λοιπόν σε ένα κράτος μέρος και εργάζονται σε ένα άλλο. Όταν αυτοί οι άνθρωποι ε, μείνουν άνεργοι, θα πρέπει να λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας από τη χώρα όπου εργαζόταν και όπου πληρώνουν τις φορές τους. Εφόσον βεβαίως έχουν εργαστεί εκεί για τουλάχιστον ένα έτος αυτό είναι ένα πιο δίκαιο και πιο απλό σύστημα από αυτό που ισχύει τώρα και τέλος σε ό,τι αφορά τα επιδόματα ανεργίας θεωρούμε ότι πρέπει κάποιος να έχει εργαστεί τουλάχιστον τρεις μήνες σε ένα άλλο κράτος μέλος πριν ζητήσουν να ληφθούν υπόψη περίοδος προηγούμενης ασφάλισης για ένα νέο επίδομα ανεργίας για να μπορέσουν να προστεθούν δηλαδή οι περίοδοι ε, κατά την οποία ήταν ασφαλισμένο ε, και εργαζόταν στο ένα κράτο και στο άλλο. Το δεύτερο σκέλο τη πρότασή μα έχει να κάνει με έναν κοινό ορισμό των μακροπρόθεσμων ωφελημάτων περίθαλψης ε, πρέπει να γίνει σαφέστερο το, το τι συμβαίνει με τα ωφελήματα αυτά ε, σε διασυνοριακές περιπτώσεις και τι δικαιούται τελικά ένας πολίτης όταν ε, μετακομίσει σε μια άλλη χώρα. Το τρίτο σκέλος έχει να κάνει με την πρόσβαση των ανθρώπων που δεν είναι οικονομικά ενεργοί σε κοινωνικά επιδόματα. Ε, θα έχετε ακούσει κι εσείς ότι πολλά κράτη-μέλη αμφισβητούν τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων κάποιος έχει πρόσβαση στο, σε, σε ωφελήματα πρόνοια, σε επιδόματα. Ε, αυτά συχνά έχουν να κάνουν με παρανοήσεις σε σχέση με τους υπάρχοντες κανόνες, αλλά δεν μπορούμε και να τα γνωρίσουμε. Δεν μπορούμε να χάσουμε τη μάχη της κοινή γνώμης ό,τι αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία. Πρέπει να εξηγήσουμε λοιπόν ποιοι είναι αυτοί οι κανόνες, γιατί αυτοί οι κανόνες είναι δίκαιοι και πώς εφαρμόζονται. Στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουμε κωδικοποιήσει μια σειρά από σημαντικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που καταλήγουν στο ότι η ελεύθερη κυκλοφορία δεν σημαίνει ότι υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε κοινωνικά επιδόματα χωρίς όρους σε άλλες χώρες. Μπορεί να έχει κάποιος πρόσβαση σε τέτοια επιδόματα και σε περίπτωση με βάση ε, ε, ένα, μια νόμιμη άδεια παραμονής. Πρέπει δηλαδή να έχει επαρκή εισοδήματα και να έχει κάλυψη ασφαλιστική. Αυτό ισχύει και τώρα, αλλά η νέα πρόταση το καθιστά πιο σαφές. Επίσης καθορίζει το ποιους αφορά. Αφορά δηλαδή ανθρώπους που δεν εργάζονται και που δεν αναζητούν εργασία. Επίσης ευθυγραμμίζουμε την ορολογία ε, σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση και με την απόσπαση εργαζομένων. Αλλά δεν αλλάζουμε τους κανόνες κοινωνικής ασφάλισης για τους αποσπασμένους εργαζόμενους. Οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι παραμένουν ε, συνδεδεμένοι με τα συστήματα κοινωνική ασφάλιση τη χώρα προέλευσή του, εφόσον έχουν αποσπαστεί για λιγότερο από 24 μήνε. Η πρότασή μα λοιπόν προβλέπει σαφέστερε διαδικασίε για τι εθνικέ αρχέ για να μπορούν να γνωρίζουν καλύτερα και πιο εύκολα ποιο είναι το καθεστώ ε, των, προσώπων που φτάνουν στην χώρα του, να αποφύγουμε έτσι τι καταχρήσει είχαμε αυτή την ομάδα ad hoc της Διοικητικής Επιτροπής που μας βοήθησε για να το πετύχουμε αυτό. Τώρα τι δεν συμπεριλαμβάνει η πρόταση. Η Κομισιόν αποφάσισε να μην προτείνει τροποποίηση στους κανόνες σε ό,τι αφορά την εξαγωγή των επιδομάτων για παιδιά. Σε κάποια κράτη-μέλη υπήρξαν σημαντικές αντιδράσεις από την κοινή γνώμη τα στοιχεία που έχουν προκύψει και σε ό,τι αφορά το οικονομικό αντίκτυπο και σε ό,τι αφορά ε, την επιβάρυνση την ε, διοικητική ε, δείχνουν ότι δεν δικαιολογείται να αλλάξουμε κάτι εδώ. Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να λέει από τη μία ότι τα πρόσωπα μπορούν να έχουν δικαίωμα για την ίδια αμοιβή, σε ό,τι αφορά την ίδια δουλειά στο ίδιο μέρος και ταυτόχρονα να δέχονται άνθρωποι οι οποίοι συνεισφέρουν στα ίδια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης με το ίδιο πόσο να την χάνουν ε, άλλου επίπεδου ε, επιδομάτων ε, για τα παιδιά τους. Αυτό είναι θέμα ε, δί, δίκαιης και ίσης μεταχείρισης. Υπήρξε βεβαίως μια συμφωνία στο τεφόρο Βασίλειο πέρυσι ε, στη διαπραγμάτευση ε, σε μια ελπίδα, με την ελπίδα μάλλον ότι το βασίλειο θα παρέμεινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν μια δύσκολη συμφωνία τότε και οδηγηθήκαμε σε έναν διακανονισμό ο οποίο είχε διαφορετική ε, κατεύθυνση. Βεβαίω υπήρχε και μια ρήτρα που έλεγε ότι αυτή η συμφωνία, αυτό ο διακανονισμό ε, δεν ισχύει με βάση το αρνητικό αποτέλεσμα ε, της, ε, του δημοψηφίσματος. Οι προτινόμενες αλλαγές λοιπόν οδηγούν σε περισσότερη διαφάνεια, νομική ασφάλεια και ε, δικαιοσύνη για τους εργοδότες, τους φορολογούμενους, τις δημόσιες αρχές θα διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία αυτό το σύστημα και θα έχουν τα κράτη-μέλη περισσότερα εργαλεία για να αποφεύγουμε τις καταχρήσεις υπήρξε συνεχής διάλογος και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με τα κράτη-μέλη καθώς και με άλλους εμπλεκομένους φορείς. Έχουμε ακούσει τις παρατηρήσεις τους, τις προτάσεις τους και είμαι διατεθειμένη να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου έτσι ώστε να προχωρήσουμε ομαλά και γρήγορα σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο φάκελο που αποτελεί προτεραιότητα της συμφωνίας ε, των τριών θεσμών για το 2017. Είμαι στη διάθεσή σας για να συνεχιστεί αυτή η ανταλλαγή απόψεων μαζί σα, ε, Τις απόψεις σα τι εκτιμώ ιδιαίτερα. Ελπίζω να έχουμε ε, αγαστή συνεργασία και αυτό να οδηγήσει στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και για την Ευρώπη και για τους συμπολίτε μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχει και χρόνο για ερωτήσει. Εγώ είμαι στη διάθεσή σα. Πολύ ωραία. Έχουμε πολλές ερωτήσεις. Και θα δώσω το λόγο στον εισηγητή και τους σκιώδης εισηγητές. Θα σας παρακαλέσω να περιοριστείτε όμως στα δύο λεπτά ο καθένας για να αφήσουμε ένα σύντομο περιθώριο για απαντήσεις. Ο κύριος Μπάλαστ λοιπόν, εισηγητής. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, ευχαριστώ πολύ για την τοποθέτησή σας και τη σαφήνεια. Στο θέμα αυτό του συντονισμού των κοινωνικών πολιτικών επιλέξατε μια σωστή μεθοδολογία με νέες προτάσεις, σαφείς, και τώρα πρέπει το Κοινοβούλιο να επιληφθεί και να τη συζητήσει. Δεν νομίζω ότι σήμερα ρόλος μου πρέπει να είναι να αρχίσω να δίνω κατευθύνσεις. Αργότερα, όταν θα έχω μελετήσει, μαζί βέβαια με τους σκιώδεις εισηγητές, το σύνολο των προτάσεων. Ίσως όμως θα μπορούσα να δώσω κάποια μεθοδολογικά στοιχεία και σημεία στα οποία πρέπει να επαγρυπνούμε. Ως προς την επαγρύπνηση λοιπόν, εσείς αναφερθήκατε στο Brexit κύριε Επίτροπε, που θα πρέπει να αναλυθεί σε όλες τις πιθανές συνέπειές του, κυρίως για την μεταβατική περίοδο, από τη στιγμή δηλαδή της απόφασης του Βρετανικού, της Βρετανικής κυβέρνησης και της υλοποίησης της αποχώρησης Βρετανίας, πώς το νέο αυτό δεδομένο στην τωρινή χρονική περίοδο μπορεί να ενσωματωθεί στη δουλειά που κάνουμε σε σχέση με την κοινωνική ασφάλιση και νομοθεσία. Για δεύτερο στοιχείο επαγρύπνησης, είναι πολύ σημαντικό πιστεύω το ότι έγινε ε, διαβούλευση με τα κράτη-μέλη, αλλά πιστεύω και οι κοινωνικοί εταίροι, εργοδότες ή εργαζόμενοι με τα συνδικάτα τους, θα πρέπει και αυτοί σήμερα ήδη να εμπλακούν στη συζήτηση ώστε ήδη από τώρα να είναι γνωστές ε, οι διεκδικήσεις τους, ε, τα σημεία στα οποία βλέπουν κινδύνους, ε, οι απαιτήσει τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα κάνουμε οτιδήποτε ζητήσουν, αλλά πρέπει να γίνει βάθος συζήτηση και με τους εκπροσώπους των εργαζομένων στα θέματα αυτά. Και ολοκληρώνω, Πρόεδρε, λέγοντας ότι στο θέμα των προτάσεων που έχουν διατυπωθεί. Θετικό είναι το ότι εν γέν και μπορούμε να τις υποστηρίξουμε, αλλά θα πρέπει να τις εμβαθύνουμε και να τις συμπληρώσουμε. Και εγώ προσωπικώς προσβλέπω σε έναν έγκαιρο διάλογο με τους και πριν την καταθέση των προτασών μας. Η Πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Σούλτσα. Δύο λεπτά. Κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστώ που ήρθατε στην Επιτροπή μας και να σας πω πως αυτά τα οποία παρουσίασε η Κομισιόν είναι μια πολύ καλή βάση επί της οποίας μπορούμε να εργαστούμε και στόχος μας θα πρέπει να είναι να διευκολύνουμε την ελεύθερη μετακίνηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα ήθελα όμως επί τη ευκαιρία να αναφερθώ σε δύο-τρία σημεία που αναφέρατε και εσείς. Το πρώτο είναι το θέμα των επιδομάτων για παιδιά, για αλλοδαπούς πολίτες της ε, Ένωσης ε, και, την, και εξαγωγή αυτών των επιδομάτων. Πρόκειται για τελείως διαφορετικά νούμερα από αυτά τα οποία είπατε που μιλήσατε για μόνο 1% και για εμένα. Αν και το αναφέρατε δεν μπορώ να αντιληφθώ πως ε, προσφέρθηκε κάτι στους ε, Βρετανούς ε, και απορρίφθηκε. Γίνεται αυτή η συζήτηση στην ε, Επιτροπή μας, ανοιχτή συζήτηση και δεν πρέπει να την παραμελήσουμε. Δεύτερον, το θέμα της απόφασης ε, του ΔΕΚ που δικαίωσε τον αποκλεισμό ορισμένων κατηγοριών αλλοδαπών από κοινωνικά επιδόματα και πώς σκοπεύει να το κωδικοποιήσει αυτό η Κομισιόν. Θα θέλαμε κάποια σαφήνεια εδώ πέρα. Και το τρίτο θέμα είναι τα επιδόματα ανεργίας και η εξαγωγή τους ε, και λέτε από τρεις σε έξι μήνες. Γιατί έξι μήνες και γιατί όχι όλο το διάστημα είναι η ερώτηση. Αυτά δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο στον χρόνο που έχω. Σας ευχαριστώ κυρία Χάρκιν για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την Επίτροπο. Νομίζω πως αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει αυτή η πρόταση είναι να καταστήσει τη στενότερη τη σχέση μεταξύ το που πληρώνονται εισφορές και που λαμβάνονται επιδόματα και να υπάρχει μία ίσο κατανομή του βάρους μεταξύ των κρατών μελών. Και η πρόταση αυτή νομίζω πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Κάποιες ερωτήσεις. Αυτό το οποίο είπε ο κ. Σούλτς για αυτό το οποίο προσφέρθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο κάποια στιγμή, το οποίο όμως ε, μετά αποσύρθηκε και βεβαίω έχουμε μια γενική εικόνα. Είπατε το νούμερο, δεν το θυμάμαι. Ένα 2% κάτι τέτοιο. Νομίζω πως ε, μια ανάλυση ανακράτος μέλος θα ήταν πολύ χρήσιμη και ε, θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε κάτι τέτοιο γιατί το βάρος σε κάποια κράτη-μέλη μπορεί να είναι πολύ μεγάλο, ειδικά αν είναι μικρές φορές. Και ίσως είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε. Ε, είναι όμως κάτι το οποίο χρειαζόμαστε. Επίσης, ήθελα να κάνω μια ερώτηση για μια απάντηση που δώσατε σε μια ερώτηση για τον ε, εξαρτώνται τα κοινωνικά υπεδόματα» από την ε, άδεια διαμονή στο την απόφαση 308-2014 Κομισιόν εναντίον Ηνωμένου Βασιλείου και αναγνωρίσατε ότι πρόκειται για μια σημαντική διευκρίνηση στο δικαίωμα πρόσβασης κοινωνικών επιδομάτων και η απόφαση επιβεβαίωσε πως υπάρχει μεγάλη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών και ότι η Κομισιόν ε, αναλύει την απόφαση για να βγάλει τα συμπερασματά της. Δηλαδή η απόφαση ήταν ότι το να εξαρτώνται τα κοινωνικά επιδόματα από το, το δικαίωμα μόνιμης κατοικίας δεν ήταν διακριτική μεταχείριση και δεν απαγορεύεται. Θα ήθελα το σχόλιο σας από αυτού και πώς ε, το έχετε ενσωματώσει αυτό στην πρόταση την οποία έχουμε τώρα μπροστά μας. Γιατί ένα από αυτά τα οποία μας λέτε είναι ότι βασίζεστε στην απόφαση του ΔΕΚ. Σε ευχαριστώ. Τζιν Λάμπερτ από τους Πράσινους έχετε τον λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Υπάρχουν κάποια πράγματα στην πρόταση αυτή θετικά Προσωπικά είμαι πολύ χαρούμενοι που δεν κάνατε αλλαγές για τα επιδόματα τέκνων. Αυτό ήταν πάντα ένα ζήτημα πολιτικό παρά κάτι το οποίο αφορούσε την ισότητα στο χώρο εργασίας. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που δεν ε, περιελήφθη στην πρόταση αυτή. Για την επέκταση την περίοδου κατά την οποία μπορεί ο κόσμος να ψάχνει δουλειά. Γενικώ το στηρίζει η ομάδα μου και για το θέμα των τριών μηνών πριν να μπορεί κάποιος να λάβει επίδομα αλλού. Πρέπει να δούμε πώς το ορίζουμε, γιατί για πολύ κόσμο αυτοί οι πρώτοι μήνες δουλειά μπορεί να είναι μια δουλειά προσωρινή ή επισφαλής και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Επίσης, στηρίζουμε το ότι όταν κοιτάμε την πλευρά της κοινωνικής ασφάλισης δεν προσπαθούμε να λύσουμε προβλήματα απόσπασης εργαζομένων μέσω του μηχανισμού κοινωνικής ασφάλισης. Ειδικά όταν ξέρουμε ότι έχουμε τόσα πολλά άτομα, από άτομα που πηγαίνουν ένα-δύο μέρες μέχρι άτομα τα οποία ε, αποσπάνονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τώρα, για το θέμα της ε, μόνιμης κατοικίας και της πρόσβασης σε επιδόματα είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε πολύ στενά έτσι ώστε να μην αποκλείονται κάποιοι από την μόνιμη κατοικία λόγω ασαφών ή λάθος αποφάσεων των κρατών μελών που θα δημιουργούν μετά δυσκολίες στα εν λόγω άτομα. Και επειδή βεβαίως μιλάμε για συντονισμό κοινωνικής ασφάλειας υπάρχει πάντα ένα πρόβλημα με τα μέτρα γέφυρα όταν τα άτομα πηγαίνουν από το ένα σύστημα στο άλλο. Πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε τα άτομα για να μην χάνονται ε, στο μεσοδιάστημα, θα έλεγα, μεταξύ δύο κρατών μελών. Ευχαριστώ. Κυρία Χέλγκα Στέβενς, μόλις έφτασε. Έχετε δύο λεπτά. repeat, we are, we are... Το επαναλαμβάνω. Θα σας παρακαλέσουμε να, τηρήσουμε, να τηρήσετε το χρόνο σας δύο λεπτά. Γιατί έχουμε πολλούς ανθρώπους που ενδιαφέρονται να τυπώσουν ερωτήσεις και θέλουμε να ακούσουμε την ε, Επίτροπο της απαντήσεις της. Έχετε το λόγο κυρία Στέβανση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Με συγχωρείτε για την καθυστέρησή μου να στην Επιτροπή Λίμπε. Είναι δύσκολη ημέρα ε, για μένα σήμερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Τάισεν για τις προσπάθειές της που προσπαθεί να κάνει κατά του τουρισμού των επιδομάτων και την όλη αυτή συζήτηση για τον σχετικό κανονισμό. Είναι λοιπόν ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολύ το κόμμα μου και θεωρούμε πως είναι κάτι το οποίο υποσκάπτει την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών και των φορολογουμένων οι οποίοι βλέπουν ότι πληρώνουν φόρους ε, και βλέπουν ότι ε, αυτοί καταλήγουν συχνά σε άτομα που έρχονται από άλλες χώρες χωρίς να έχουν εισφέρει ποτέ στο σύστημα κοινωνικής ε, ασφάλισης. Αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται να δουλέψουν είναι βεβαίως ε, καλοδεχούμενοι, αλλά ε, όχι ε, εις βάρος, να έρχονται άνθρωποι εις των εργαζομένων. Λοιπόν, κάποιος ο οποίος έρχεται λοιπόν για να εργαστεί είναι όπως είπα ευπρόσδεκτος και θα πρέπει όμως να εισφέρει πρώτα στο σύστημα πριν μπορέσει να εκμεταλλευτεί τα θετικά του και θα πρέπει όπως είπαμε να αποφύγουμε το κοινωνικό ντάμπινγκ μέσω της απόσπασης εργαζομένων γιατί θα πρέπει, όπως είπαμε, η απόσπαση θα πρέπει να είναι το πολύ δύο χρόνια σε μια άλλη χώρα χωρίς να πληρώνει κανείς ε, εισφορές στη χώρα την οποία εργάζεται. Γιατί τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, συγκεκριμένα στη δική μου τη χώρα, η Βέλγοι είναι πάρα πολύ ακριβοί για να απασχοληθούν στο Βέλγιο τελικά, γιατί υπάρχουν άλλοι οι οποίοι πληρώνουν σε άλλη χώρα χαμηλότερες κοινωνικές ε, εισφορές. Ε, ε, οπότε όταν λέμε ίδια δουλειά, ίδια πληρωμή για ίδια εργασία, ε, αυτό περιλαμβάνει βεβαίως ε, και τις ε, κοινωνικές εισφορές και βεβαίως θα πρέπει ακριβώς στους επικίνδυνους τομείς να περιορίσουμε την διάρκεια της απόσπασης τους έξι μήνες και τα κράτη-μέλη να αποφασίσουν μόνα τους ποιοι είναι οι επικίνδυνοι τομείς για κοινωνικό ντάμπινγκ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα σε εμά είναι η οικοδομή παραδείγματος χάρη, όπου έχουμε αθέμητο ανταγωνισμό. Σας, σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Στίβενς. Τώρα θα παρακαλέσω την Επίτροπο να λάβει το λόγο για να απαντήσει στις ε, ερωτήσεις που έχουμε μέχρι τώρα ακούσει και ελπίζω ότι θα έχουμε περιθώριο για, μερικές, για μια σειρά ακόμα ερωτοπαντήσεων. Α, η Γκουε. Είχα άλλο όνομα. Καλώς, ναι. Σας δίνω το λόγο λοιπόν εκ μέρους της Γκουε, κυρία Λόπες Φερμέρο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστώ την Επίτροπο ε, Τάισεν. Ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης είναι ένα θέμα ε, αδιαφυσβήτητα σημαντικό. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, όπως λέει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχουν τουλάχιστον 11 εκατομμύρια Ευρωπαίοι που ζουν σε μια χώρα άλλη από τη χώρα προέλευσή του. Και υπάρχουν και βεβαίω εκατομμύρια εργαζόμενοι αποσπασμένοι. 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενοι επίση εργάζονται διασυνοριακά. Αυτό είναι μια εικόνα τη στιγμή. Αλλά καθ' όλη τη διάρκεια τη ε, ε, ζωή του είναι εκατομμύρια οι πολίτε οι οποίοι εργάζονται και συνεισφέρουν σε διάφορε χώρε στην Ευρώπη. Υπάρχουν πολλά σημεία που θα υποβάλουμε τροπολογίε. Ε, η πρότασή σας πάντως πάει προς τη σωστή κατεύθυνση. Η φορητότητα των επιδομάτων ανεργίας παραδείγματος χάρη ή ε, τα οικογενειακά επιδόματα. Πέρα όμως από τις θετικές αυτές πτυχές υπάρχουν δύο θεμελιώδη ζητήματα όπου έχουμε σημαντικά κενά. Οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι και η προστασία του θεμελιώδη δικαιώματος της κινητικότητας των εργαζομένων. Και θέλω να σας υποβάλω δύο ερωτήματα. Πρώτον, γιατί επελέξατε να πάτε στους 24 μήνες ό,τι αφορά τις αποσπάσεις, όταν οι περισσότερες αποσπάσεις διαρκούν 4 με 6 μήνες. Ουσιαστικά αρνείστε να χορηγήσετε κοινωνική, κοινωνική ασφάλιση σε αυτούς τους αποσπασμένους ε, εργαζόμενους. Αυτό δεν δίνει έναν πυρήνα δικαιωμάτων στους υποσπασμένους εργαζόμενους για να αποφύγουμε το κοινωνικό ντάμπινγκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το δεύτερο, ίσως και πιο σοβαρό, δεν αιτιολογείται το να χάνουν δικαιώματα οι άνεργοι. Διότι αυτό, το να φέρει κάποιες δικαιώματα, είναι σαν να φέρει την ίδια την ηθαγένεια ενός πολίτη. Μιλάω για τους ανθρώπους οι οποίοι πάνε σε ένα άλλο κράτο μέλο να χάνουν τη δουλειά του. Ε, γίνεται διαπραγμάτευση με τον Ηνωμένο Βασίλειο για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, αλλά στο Βέλγιο υπάρχουν Ιταλοί και Ισπανοί πολίτε ε, οι οποίοι ε, εκδιώκονται από τη χώρα. Ευχαριστώ. Και τώρα κύριε Τάισον. Για να ακούσουμε απαντήσεις σαφείς και σύντομε για να έχουν το χρόνο και άλλοι συναδελφοί να δείτε πώ είναι τι ερωτήσεις τους. Ευχαριστώ ε, στα άλλα Ολλανδικά. Πρώτα απ' όλα, καλή επιτυχία στον εισηγητή και ελπίζω να λειτουργήσει η προσέγγιση σας. Δεύτερον, υπήρχε το ερώτημα για το Brexit. Κοιτάξτε, οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν με βάση το άρθρο 5, αλλά όσο δεν έχουν ξεκινήσει και όσο δεν έχουν ολοκληρωθεί, εξακολουθεί να είναι μέλος της Ένωσης ε, το Ηνωμένο Βασίλειο και έχει όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις ε, των άλλων κρατών μελών και οι πολίτες ε, επίσης έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις. Αν όταν υπάρξει αυτή η συμφωνία αποχώρησης, αυτή η συμφωνία θα ρυθμίζει και τα σχετικά, αλλά μέχρι να αποφασιστεί κάτι τέτοιο ισχύουν ε, τα προηγούμενα. Για το επίδομα τέκνων. Γιατί δεν κάνουμε κάποια πρόταση για να τροποποιηθεί ανάλογα με το επίπεδο της χώρας που μένουν τα παιδιά, αν μένουν σε άλλη χώρα από τους εργαζόμενους γονείς ή γονέα. Κοιτάξτε να δούμε περί τίνος ε, πρόκειται, είδαμε περί τίνος πρόκειται και για τι αριθμούς μιλάμε, για πόσα άτομα μιλάμε. Είναι λιγότερο από 1% τα παιδιά που ζουν σε άλλη χώρα από τον εργαζόμενο γονιό. Δηλαδή, αν προσαρμόζαμε δε το συγκεκριμένο επίδομα θα ήταν λιγότερο από το 1% του συνολικού κόστους. Λοιπόν, αν ρωτούσαμε τα κράτη-μέλη εάν θα ήθελαν αυτή την ευκαιρία θα το προσάρμοζαν σε κάθε ένα από τα άλλα 27 κράτη-μέλη και θα έπρεπε να υπάρχει και τακτική προσαρμογή. Μπορεί επίσης να υπάρχει προσαρμογή προς τα κάτω αλλά και προς τα πάνω. Έτσι, αν ε, το κόστος ζωής είναι ακριβότερο από εκεί που εργάζεται ο γονιός, ε, θα συνέβαινε και κάτι τέτοιο. Και θα, θα ίσχυε επίσης το ίδιο και για τους ίδιους τους πολίτες του κράτους που ε, θα έκανε κάτι τέτοιο. Αν ήταν σε άλλη χώρα. Έτσι, γιατί δεν γίνεται να υπάρχει διακριτική μεταχείριση με βάση την εθνικότητα. Αλλά το σημαντικότερο για εμάς είπαμε ότι θέλουμε ξεκάθαρους ε, κανόνες που να εφαρμόζονται εύκολα, δεν θεωρούμε ότι εφαρμόζεται εύκολα κάτι τέτοιο και είπαμε στην ε, πρότασή μας για τους αποσπασμένους ότι για ίδια εργασία στο ίδιο μέρος θα πρέπει να υπάρχει ίδια πληρωμή ε, δεν μας φαίνεται πολύ δικαιολογημένο μετά να πούμε ότι εξαρτάται από το που πληρώνει κανείς ή το που είναι τα παιδιά του. Λοιπόν, αν κάποιος άλλος ε, δουλεύει στο... και πληρώνει τις ίδιες φορές στην ίδια χώρα, πρέπει να μπορεί να παίρνει και τα ίδια επιδόματα. Νομίζω είναι λογικό και δίκαιο. Και βεβαίως θα χρειαζόταν και αλλαγή νομοθεσίας. Αυτά λοιπόν για το επιδόματο το Υπήρχε το ερώτημα για το επίδομα ανεργίας, γιατί δεν μπορεί να μεταφέρεται ε, και αν μπορεί να μεταφέρεται από κάποιον ο οποίος πάει να αναζητήσει δουλειά σε μια άλλη χώρα. και από τρίμηνο ε, να γίνει εξάμηνο στο μέλλον και ρώτησε κάποιος γιατί να μην είναι αόριστη η διάρκεια. Γιατί γνωρίζουμε ότι εντάξει, λογικό είναι ε, να υπάρχει ένα εύλογο διάστημα εντός του οποίου μπορεί κανείς να πει ότι αναζητεί δουλειά. Νομίζω ότι έξι μήνες είναι λογικό. Και καλό είναι να μπορεί κανείς να μεταφέρει το επίδομα ανεργία σε μια άλλη χώρα για να αναζητήσει εκεί πέρα δουλειά. Έχει περισσότερες πιθανότητες να βρει. Μετά, το ερώτημα για την ομολογία την οποία δεν έχουμε ακόμα κωδικοποιήσει στην πρόταση αυτή. Ποιο? Ναι, η υπόθεση Αλεμάνοβιτς για κοινωνική προστασία. Δεν είναι θέμα κοινωνικής ασφάλισης ε, στρίκτου σένσου και δεν ε, μπορεί να ρυθμιστεί άρα με αυτήν την ε, οδηγία η υπόθεση Κομισιών αντίον Ηνωμένου Βασιλείου πράγματι αφορούσε κοινωνική ασφάλιση και θα κωδικοποιηθεί. Και σημαίνει ότι μπορεί πράγματι ένα κράτος μέλος να θέσει ως προϋπόθεση πρόσβασης ε, στο σύστημα το δικαίωμα μόνιμης κατοικίας. Δηλαδή μπορεί να αρνηθεί σε κάποιους ε, την ε, πρόσβαση και αφορά τα, ε, άτομα τα οποία δεν είναι οικονομικά ένεργα, ε, ούτε εργαζόμενους ούτε όσοι αναζητούν εργασία. Και μετά ήταν το ερώτημα της κυρίας ε, Στίβενς που έκανε σύνδεση μεταξύ του συντονισμού και των αποσπασμένων εργαζομένων και γιατί η περίοδος των δύο ετών που δίνει την ευκαιρία να πληρώνουν κοινωνικές φορές στη χώρα στην οποία έχουν τη σύμβαση εργασίας. Γιατί πρώτον, και εδώ πέρα δεν θέλουμε να κάνουμε υπερβολικές ε, γραφειοκρατικές ε, ρυθμίσεις. Ε. Δηλαδή αν έπρεπε κάθε φορά για δύο μήνες απόσπαση να αλλάζει σύστημα κοινωνικής ασφάλισης θα ήταν πάρα πολύ δύσκολα και περίπλοκα τα πράγματα και θα έπρεπε κανείς μετά να κάνει να συμπληρώσει ένα παζλ ολόκληρο για να μαζέψει τις ε, εισφορές του από εδώ και από εκεί, από διάφορα συστήματα. Αλλά κυρίως γιατί θέλουμε να διατηρήσουμε τα δύο έτη, γιατί αν το κάνουμε πολύ σύντομο τελικά θα περιορίσουμε την ελεύθερη κυκλοφορία. Και δεν το θέλουμε. Θέλουμε να την διευκολύνουμε, να έχουμε τις τέσσερις ελευθερίες κοινή αγοράς, να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους που θέλουν να το χρησιμοποιήσουν, να καταπολεμήσουμε την κατάχρηση και να βρεθεί μια ισορροπία. Και πράγματι είναι ένα σύστημα το οποίο έχουμε και σήμερα για τους αποσπασμένους. Αλλιώς θα καταργούσαμε και την ελεύθερη διακίνηση ε, υπηρεσιών, το οποίο μετά θα δημιουργούσε πρόβλημα στην ανάπτυξη που δημιουργεί θέσεις εργασίας. Ε, τελικά έτσι δηλαδή θα καταστρέφαμε θέσεις εργασίας αντί να δημιουργήσουμε και δεν νομίζω αυτό να το θέλει κανείς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Προχωράει η ώρα. Ας ακούσουμε ερωτήσεις από συναδελφούς που δεν είναι εισήγητες ή σκιώδες. Ο κύριος Μαν, ένα λεπτό. Και ένα λεπτό η κυρία Στάινρουκ. Κύριε Μαν, ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε, αγαπητή Μαριάννα. Είναι Σαφέ ότι σε μια τέτοια πρωτοβουλία δεν είναι υποχρεωτικό να συμφωνούν όλοι. Πρέπει να συζητήσουμε τα διάφορα ζητήματα. Έχω μόνο ένα λεπτό λοιπόν στη θέση μου και θα αφήσω κάποια συγκεκριμένα σημεία εκτό, αλλά θέλω να τονίσω ιδιαίτερα τη διαφάνεια οπωσδήποτε, τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων οπωσδήποτε και ιδιαίτερα των συνδικαλιστικών σωματείων που δεν εμφανίζονται εδώ και που θα πρέπει να βρούμε μια σωστή ισορροπία για τη συμμετοχή του. Και είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε και για ισονομία, για δικαιοσύνη. Βλέπουμε να υπάρχει μία κατεύθυνση που έχουν πάρει τώρα τα κράτη-μέλη ε, από διάρθρωση των κοινωνικών συστημάτων που δεν πρέπει όμως να αποτελέσει και πηγή τροφοδότησης των επιχειρημάτων των λαϊκιστών. Δεν μπορούμε να λέμε ότι ε, αφήνουμε τα κοινωνικά συστήματα να καταρρεύσουν και μετά δεν μπορούμε να, τα, ε, να καλύψουμε τις ανάγκες των ανθρώπων. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έχουμε μία προσέγγιση η οποία θα διατηρήσει τις βασικές αξίες. Ευχαριστώ. Τώρα λεπτό προφανώς δεν αρκούσε. Κυρία Στάινρουκ, εν όλο η πρόταση της Επιτροπής μου φαίνεται ευπρόσδεκτη και για το επίδομα ανεργίας και για την υποστήριξη ε, του εισοδήματος των οικογενειών μικρά παιδιά. Η αναπροσαρμογή είπατε μπορεί να οδηγεί σε προβλήματα σχέση με τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών κρατών. Καλό θα είναι να μην καμφθούμε ενώπιον των λαϊκιστών και να μην εμποδίσουμε την ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προφανώς έχει αναφερθεί και έχει λάβει υπόψη την τελευταία απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικοστηρίου, αν και εγώ διαφωνώ στην ε, αξιολόγησή της και στην ανάλυση της. Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι δεν μπορεί αδίποτε διοικητική παρέμβαση της Επιτροπής να αντικαταστήσει τον ε, κοινωνικό διάλογο. Η απόσπαση επίσης Καλό θα είναι να μην αφήσουμε ασαφείς τις έννοιες ε, στο κανονισμό 883. Είναι ασαφείς ακόμη πολλές έννοιες και θα πρέπει, επί παραδείγματι στο άρθρο 12, όπου αναφέρεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον αποσπασμένο εργαζόμενο, αφενός αφετέρου στον αποσταλέντα εργαζόμενο. Μέσα στο ίδιο άρθρο έχει δύο φορές διαφορετικές έννοιες και άρα χρειάζονται και διαφορετικοί ορισμοί για να ξέρουμε τι λέμε γιατί είναι πολύ περίπλοκη η κατάσταση. Κύριε Τάισον. Τώρα έχετε το χρόνο στη διάθεσή σας για να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι η σημαντικότερη αντίδραση των ε, δύο τελευταίων συναδέλφων ε, έχει να κάνει με την εμπλοκή των κοινωνικών τέρων. Η πρόταση αυτή δεν βασίζεται στο άρθρο 153, το οποίο κανονικά αφορά την διαβούλευση των κοινωνικών εταίρων, αλλά βεβαίως ενημερώνονται οι κοινωνικοί εταίροι τακτικά μονίμως ε, πριν ε, εκπονήσουμε μια πρόταση. Δεν την κάναμε στον για πύργο του Μπερλεμόν απομονωμένη. Βεβαίως υπήρχε διαβούλευση με τους ε, κοινωνικούς εταίρους ε, από την ε, τριμερή διαβούλευση. Και ακούσαμε τις παρατηρήσεις τους και αν υπάρχουν κάποια πράγματα στους ορισμούς που δεν είναι σωστά βασιζόμαστε στην ε, σοφία του Κοινοβουλίου να υποβάλει τις σωστές ε, τροπολογίες και να τα διορθώσει. Νομίζω το σημαντικότερο μήνυμα, κυρία Πρόεδρε, είναι πως ε, ελπίζουμε να κλείσει ο πρώτος γύρος με τα πράγματα αυτά τα οποία πρέπει να αλλάξουν όπως είπαμε στον κανονισμό. Υπάρχουν αλλαγές ε, στην οικονομία, στον τρόπο εργασίας ε, και να δούμε πώς θα μπορέσουμε επίσης να ενσωματώσουμε την νομολογία και να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε κάποιες παρεξηγήσεις ε, για να δημιουργήσουμε ακριβώς ευκαιρίες και να μπορεί ο κόσμος να διαβάζει με λόγια ξεκάθαρα το τι συμβαίνει στην ε, περίπτωσή του. Αυτά και σας ευχαριστώ για την πρώτη αυτή θετική ανταλλαγή απόψεων και ελπίζω να αναπτυχθεί μια καλή δυναμική στο Κοινοβούλιο και να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό το οποίο και οι τους πολίτες. Σας ευχαριστώ που μας προσφέρετε αυτή την ευκαιρία και είστε βέβαια ευπρόσδεκτοι όποτε θέλετε στην Επιτροπή μας. Έχουμε πάρα πολλά θέματα πάντοτε να, σας, να συζητήσουμε μαζί σας. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν και σας ξαναπεριμένουμε. Λοιπόν, προτείνω να ξαναρχίσουμε. Έχουμε τώρα ένα εργαστήριο που έχουν ετοιμάσει οι υπηρεσίες μας για την εγγύηση, για την νεολαία και την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Και έτσι θα ακούσουμε τους εμπειρογνώμονές μας και θα προβούμε σε ανταλλαγή απόψεων μαζί τους. Δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίσω τη σημασία της δουλειάς αυτής, της εγγύησης για την νεολαία, της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, ιδιαίτερα το τεράστιο πρόβλημα, τη μάστιγα της ανεργίας των νέων που καθημερινά διαπιστώνουμε, μια σειρά από μέτρα έχουν εισαχθεί. Σημειώνω ότι έχουμε και έγγραφα εδώ. Μπορείτε αποχωρώντας να τα πάρετε μαζί σας. Και συζητούμε πρώτα τις επενδύσεις για την νεολαία και το ρόλο των εγγυήσεων για την νεολαία. Και δίνω το λόγο στον κύριο Τάμας Βακνάη από τη Γενική Διεύθυνση Επασχόλησης Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις εγγύησεις για την νεολαία. Κύριε Βαρνάη, ευχαριστώντα σας για την ε, παρουσία εδώ, σας καλώ να μας παρουσιάσετε τον απολογισμό των τριών τελευταίων ετών, των τριών ετών λειτουργίας των εγγύησεων για την νεολαία και βέβαια προτάσεις για τη λειτουργία τους και για την βιωσιμότητά τους. Έχετε 15 λεπτά στη διάθεσή σας. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και καλησπέρα σας. Θα ξεκινήσω την παρουσίαση παρουσιάζοντας ε, τη γραμμή του χρόνου. Πότε ξεκίνησε η εγγύηση για την νεολαία και που βρίσκεται σε σχέση με την κίνησή της. Έχουμε λοιπόν ως σημείο κίνηση τη σύσταση του Συμβουλίου τον Απρίλιο του 2013 για την εγγύηση για την νεολαία. Έως το τέλος του έτους είχαν αρχίσει να αποστέλουν τα σχέδια υλοποίηση στα κράτη-μέλη. Άρχισαν οι συνομιλίες το πρώτο ήμιση του 2014 με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό θεωρούμε ως σημείο αφετηρίας της εγγύησης για τους νέους. Με την σύνταξη λοιπόν την κατάρτιση των σχεδίων υλοποίησης, τα κράτη-μέλη ήδη είχαν καταγράψει τις ιδέες τους για τη λειτουργία της εγγύησης για την νεολαία, το σχεδιασμό των εταιρικών σχέσεων, τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, της αγοράς εργασίας, ε, της παιδείας και το καθεξής. Από το 2014 λοιπόν και μετά έχει πάρει σάρκα και ώστα η εγγύηση για την νεολαία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει την υποστήριξή της για την υλοποίηση και σε όρους χρηματοοικονομικούς και σε όρους ε, τεχνικής υποστήριξης. Έχουμε συναφείς πρωτοβουλίες επίσης που υιοθετούνται. Ευρωπαϊκή εταιρική σχέση για μαθητεία, ε, πρακτικές εξασκήσεις στο θεματολόγιο για τις δεξιότητες και άλλα στοιχεία που ενσωματώνονται και στο ευρωπαϊκό εξάμεινο και ενδεικτικό θεματολόγιο που μας ε, χρησιμεύει ως ε, πηξίδα για να παρακολουθούμε την υλοποίηση της εγγύησης για την νεολαία. Βάσει όλων αυτών, τον Οκτώβριο του 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταθέτει την πρώτη έκθεση για την εγγύηση για την νεολαία και την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Τα στοιχεία που θα σας παρουσιάσω για την εγγύηση ε, για την νεολαία είναι βασισμένα σε αυτή την έκθεση του Οκτωβρίου 2016. Βλέπετε λοιπόν εδώ τα πρώτα και κύρια αποτελέσματα που προβάλλει η έκθεση. Καταρχάς, τα καλά νέα, ότι είναι 1,6 εκατομμύρια λιγότεροι είναι νέοι άνεργοι ε, σε σχέση με την ε, κίνηση της εγγύησεως. Λιγότεροι είναι κατά 900.000 οι οι μη καταρτισμένοι, μη εκπαιδευμένη. Αρχίζει να ενισχύεται πάλι η ανάπτυξη, η απασχόληση των νέων. 1,6 εκατομμύριο νέοι υποστηρίζονται απευθείας από την πρωτοβουλία. Και βεβαίως όλα αυτά μπορούμε να τα δούμε μέσα στους κυκλικούς παράγοντες και να τα και διαφορετικά, αλλά μπορούμε να πούμε ότι η ανεργία των νέων μειώθηκε ταχύτερα από ότι η αντίστοιχη του ενήλικου πληθυσμού. Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις επίσης ε, προς οποίες έχει δώσει όθηση η ε, εγγύηση για την νεολαία ήδη έχουν δώσει αποτελέσματα. Δεν, δεν νομίζω ότι μπορείτε να το διαβάσετε αυτό που γράφουμε στο γράφημα αυτό, γιατί είναι μικρά τα γράμματα, αλλά είναι μακροοικονομικά στοιχεία αυτά που βλέπετε, τα ποσοστά της ανεργίας των νέων, το, την, το λόγο ανεργίας των νέων, και άλλα στοιχεία από το 2008 στο 2015. Από το 2008 στο 2013 βλέπουμε μια ε, τάση επιδίνωσης σε όλα τα στοιχεία εκτός από την ε, πρώιμη αποχώρηση από το εκπαιδευτικό σύστημα ενώ από εκεί και πέρα αντιστρέφεται η τάση και παρουσιάζεται μια μικρή βελτίωση. Ωστόσο παραμένουν 6 εκατομμύρια νέοι ανεκπαίδευτοι και ε, χωρίς δεξιότητες και χωρίς απασχόληση ε, για το 2015 και αυτό παραμένει υψηλότερο από τους ε, νέους νίτς όπως λέγονται του 2008 με όλες τις πρόοδους λοιπόν που σημειώνονται πάλι μένει αρκετή δουλειά να γίνει. Συγκεκριμένα τώρα για την εγγύηση για την νεολαία. Από την ε, θέση λειτουργία των Εθνικών Προγραμμάτων Εγγύησης για την Νεολαία έχουμε 16 εκατομμύρια νέους που έχουν εγγραφεί στα συστήματα, έχουν καταχωριστεί, 10 εκατομμύρια νέοι έχουν δεχθεί πρόταση είτε για απασχόληση είτε για εκπαιδευτική εκπαιδευτικό πρόγραμμα, κατάρτιση, μαθητεία, πρακτική εξάσκηση. Και χωρίς να θέλω να σταθώ στην πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων που θα ε, καλύψει προσεχής παρουσίαση. Θέλω ιδιαίτερως να τονίσω ότι η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων σημαίνει μία για πρώτη φορά υποστήριξη των νέων νίτς, των οποίων τα ποσοστά ήταν υψηλότερα το 25%, 1,6 εκατομμύρια δηλαδή, έχουν, λάβει υποστήριξη. Οικονομική υποστήριξη και σε σχέση με την εφαρμογή τις εγγύσεις για την νεολαία, αλλά αντίστοιχα και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Έχουν προσφερθεί ποσά για την υποστήριξη των ε, εθνικών προγραμμάτων υποστήριξης ε, και εγγύηση για την νεολαία. Και εδώ έχω το κύριο μήνυμα που θέλω να σας δώσω με την παρουσίασή μου, ότι η εγγύηση για την νεολαία βεβαίως εγγυάται όλα αυτά, αλλά δεν περιορίζεται μόνο σε αυτά που αναφέραμε, γιατί επιδιώκει και μακροχρόνιες ε, αλλαγές ε, και σχεδιασμό πολιτικής που θα αποτέλεσουν τη βάση της αντίληψης αυτής για την ε, εγγύηση για την νεολαία, προσβλέπει στην εξάλληψη των φραγμών μεταξύ διαφόρων τομέων δραστηριοποίησης, αλλά ακόμη και μεταξύ εταιρικών ε, ή συνεργατικών σχέσεων μέσα στις ιδέες της κυβερνήσης, Υπουργείο Εργασίας αφενός ε, και άλλα Υπουργεία ή μεταξύ εθνικών κυβερνήσεων και μη κυβερνητικών οργανώσεων, τοπικών αρχών και λοιπόν φορέων. Και αυτή, ε, αυτό το επίτευγμα είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν. Δεύτερον, Μεταρρύθμιση σημειώνεται, μεταρρυθμίσεις σημειώνονται ιδιαίτερα στα θέματα της μαθητής και της πρακτικής εξάσκησης που έχουν τεράστιο ρόλο και συμβολή στην μετάβαση των νέων από, την, ε, από το εκπαιδευτικό σύστημα στην αγορά εργασίας. Έχουν γίνει λοιπόν αυτές οι μεταρρυθμίσεις σε ένα τρίτο των κρατών μελών σημειώνονται μεταρρυθμίσεις στο σύστημα πρακτικής εξάσκησης ώστε να έχουν την ευκαιρία να μπουν σε συστήματα πρακτικής οι νέοι. Οι υπηρεσίες του δημόσιου φορέα επίσης βελτιώνουν την στόχευση των υπηρεσιών, ιδιαίτερως εκείνων που απευθύνονται προς τους νέους. Δύο τρίτα των δημοσίων φορέων ε, ορίζουν ε, συγκεκριμένες υπηρεσίες και στόχευση στη νεολαία με έμφαση και ενίσχυση και του αντίστοιχου προσωπικού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρώιμη παρέμβαση και στην κάλυψη των μη καταχωρημένων, καταχωρισμένων ε, needs, ενθαρρύνονται δηλαδή οι νέοι που δεν, έχουν, δεν είναι σε εκπαιδευτικό σύστημα απασχόληση ή κατάρτιση να καταχωρίζονται στα συστήματα αυτά στα κράτη-μέλη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί όπως ξέρετε δεν είναι διτεθειμένοι όλοι οι νέοι να απευθυνθούν σε ένα δημόσιο φορέα για να ζητήσουν υποστήριξη. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν οι υπηρεσίες, οι δημόσιες υπηρεσίες εργασίας να μπορούν να βρουν τον τρόπο να επικοινωνήσουν μαζί τους, να τους πλησιάσουν. Έχουμε ακόμα βέβαια προκλήσεις μπροστά μας. Πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά που κάνουμε στην εγγύηση για την νεολαία και για να σας παρουσιάσω το ευρύτερο πλαίσιο. Θα ήθελα να αφερθώ στην πρόταση για την νεολαία του προηγούμενου Δεκεμβρίου που αναφερόταν σε τρεις κλάδους δράσης, απασχόληση, εκπαίδευση και κινητικότητα μαθητιακή και συμμετοχή πολύ σημαντικό βεβαίω όσον αφορά τη δική μα τη δουλειά είναι το κομμάτι που αφορά την απασχόληση και η υλοποίηση τη εγγύηση για την νεολαία. Είναι πολύ καλό βεβαίω ότι ξεκίνησε και λειτουργεί η εγγύηση για την νεολαία, αλλά πρέπει να διατηρήσει την ορμή τη, την αποτελεσματικότητα και βέβαια με την κατάλληλη χρηματοδότηση και δεσμεύσει από το ευρωπαϊκό σου και από τα εθνικά επίπεδα. Πρέπει να στραφούμε περισσότερο προς τους ε, νέους που δεν είναι σε απασχόληση, μαθητεία ή εκπαιδευτικό σύστημα που δεν έχουν κατάρτιση, γιατί ξέρουμε ότι συνήθως είναι πιο εύκολα τα πράγματα για τους νίτς που έχουν υψηλή κατάρτιση και δεξιότητες. Οι λεγόμενοι μη ενεργοί δεν ωφελούνται τόσο από την εγγύηση για την νεολαία. Επίσης, εδώ έχουμε το θέμα της εξισορρόπησης της προσφοράς. Ένα από τα ευρήματα της έκθεσης της Επιτροπής ήταν ότι η προσφορά επιτοπλίστων αφορά α, θέσεις εργασίας 70%, 13% εκπαίδευση, 4% ε, μαθητεία και το υπόλοιπο πρακτική εξάσκηση. Για να στραφούμε όμως και να πλησιάσουμε τους ε, μη ενεργούς νίτς χρειάζεται περισσότερη εκπαίδευση, μαθητεία και πρακτική εξάσκηση στην προσφορά στο πακέτο της προσφοράς των προσφερόμενων υπηρεσιών. Πρέπει να συνεχίσουμε να ενισχύουμε το θεσμικό δυναμικό και τι εταιρικέ σχέσει και τι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδο, όπω είπα, παραμένουν ακόμα κάποιε επικρίσει. Και ίσω το πιο σημαντικό ε, στοιχείο είναι αυτό που αφορά την ποιότητα τη προσφορά. Είτε είναι πολύ βραχυπρόθεσμη η προσφορά, είτε δεν είναι χρήσιμη για το νέο μακροπρόθεσμα, για να ενσωματωθεί μακροπρόθεσμα στην αγορά εργασίας μαθητείες παραδείγματι που δεν έχουν γνωστικό περιεχόμενο ή δεν εξασφαλίζουν επαρκείς ε, συνθήκες εργασίας, ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας. Πέραν αυτού βεβαίως θα σημειώσω για τη μαθητεία ότι έχουμε ένα πλαίσιο ποιότητα που προσδιορίζει την ε, μαθητεία αλλά και για την ε, πρακτική εξάσκηση. Ετοιμάζεται να προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα πλαίσιο περιεχομένου. Η ποιότητα όμως πρέπει να προωθεί ακόμη περισσότερο. Και η Επιτροπή Απασχόληση αλλά και η Επιτροπή ΙΜΚΟ θα ε, έχουν την ευκαιρία να δουν τις προτάσεις αυτές. Συνεχίζεται λοιπόν η χρηματοοικονομική υποστήριξη. Για το μέλλον σκοπεύουμε να συνεχίσουμε την υποστήριξη στο 2018 και από το Κοινωνικό Ταμείο στο 2020 η πρωτοβουλία για την απασχόληση για των νέων ξέρουμε ότι ακόμη δεν έχει προσδιοριστεί το ποσό που θα την, με το οποίο θα πρικοδοτηθεί είναι σε συζήτηση, σε επίπεδο συζητήσεων στο Κοινοβουλίο, αλλά βεβαίω όλα αυτά μπαίνουν σε ένα ευρύτερο πακέτο για την υποστήριξη τη νεολαία. Όπω είπαμε, υπάρχει το δεύτερο και το τρίτο σκέλο του πακέτου προτάσεων για την νεολαία. Το δεύτερο σκέλο αφορά την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης κινητικότητας στην ε, πρακτική εξάσκηση και το ποιοτικό πλαίσιο και επίσης ε, η αλληλεγγύη και η εταιρική σχέση με το Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών και Αλληλεγγύης που ετοιμάζει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα προσφέρει ευκαιρίες για τους νέους να προχωρήσουν και να ενσωματωθούν στην αγορά εργασία. Νομίζω ότι έχω φτάσει στο τέλος της ε, παρουσίασής μου. Πολύ σύντομα λοιπόν, γιατί ξέρω ότι δεν μπορείτε να τα διαβάζετε αυτά, ε, στην εξισορρόπηση των ε, προσφερωμένων υπηρεσιών από την εγγύηση για την νεολαία. Βλέπετε την απασχόληση η οποία κατέχει το 70% και η τελευταία τελευταία διαφάνεια γιατί θέλω να επισημάνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, υποστηρίζει και ε, περαιτέρω προτάσεις για την εγγύηση για την νεολαία. Αυτά λοιπόν ε, είναι μια απεικόνηση, μια γραφική παράσταση που αναφέρεται ακριβώς σε αυτή την ιδέα. Πολύ ευχαρίστω ε, βεβαίω να, σα να απαντήσω σε ερωτήσει μαζί με τα στοιχεία μου που σα αφήνω εδώ. Ευχαριστώ ιδιαίτερα για όλε αυτέ τι εξηγήσει. Και τώρα οι εισηγητέ για δύο λεπτά ο καθένα, Η κυρία Ρωμανάτομ. Non. Non. Sinon, M. n'est pas là. Από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Λείπει ο συνάδελφος, οπότε θα μιλήσω εγώ εκ μέρους της πολιτικής μας ομάδας. Θέλω να κάνω μια σειρά από σχόλια για την παρουσίαση. Πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία. Ε, κάποια είναι θετικά και ενθαρρυντικά, όπως η μείωση, η σαφής μείωση της ανεργίας των νέων και η σχέση μεταξύ του ευρωπαϊκού σχέδιου για τις ε, εγγυήσεις για τους νέους και των δημοσίων πολιτικών που ακολούθησαν σε εθνικό επίπεδο ε, χάρη σε αυτή την ομπρέλα της εγγύησης για τους νέους. Ε, αυτά είναι θετικά. Βεβαίως υπάρχουν και μεγάλες διαφορές κατά την εφαρμογή. κάποια στοιχεία θα πρέπει να μας ανησυχήσουν και υπάρχουν και κάποια πιο δομικά ζητήματα. Καταρχήν για το ε, ποσοστό κάλυψης. Είναι τεράστιες οι διαφορές. Σε ό,τι αφορά τώρα την ε, ομάδα ανθρώπων στους οποίους εστιάζουμε. Έχουμε 80% ε, ατόμων εγγεγραμμένων στην Αυστρία, στην Ιταλία, στην Ισπανία 10%. Στη Γαλλία πάλι 80%. με βάση την αξιολόγηση της Κομισιόν το περασμένο φθινόπωρο, έτσι. Το έχουμε εξετάσει αυτό σε βάθος. Έχουμε και κάποιες αμφιβολίες ε, γιατί σε κάποιες χώρες το ποσοστό επιτυχίας είναι υψηλότερο από ό,τι σε άλλες. Γιατί ε, μετά από έξι μήνες ρωτάμε σε κάποιες χώρες ε, ε και οι απαντήσεις είναι θετικές 71% θετικές απαντήσεις στην Ιρλανδία, 64% στην Ιταλία, στην Ισπανία 37%, στην Ουγγαρία 30%. Αυτό μας ανησυχεί. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές και σε ό,τι αφορά την κάλυψη, τους πόσους ανθρώπους καλύπτουμε και, και σε ό,τι αφορά την επιτυχία του όλου προγράμματος. Ε, μάλιστα, ευχαριστώ. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποιος άλλος από την Άλντε. Παρακαλώ συγγνώμη αν δεν πρόφερα σωστά το όνομά σας. Προσπαθήσατε όμως, προσπαθήσατε. Ε, δεν είναι, θέλω να μιλήσω εδώ και ο με τους εμπειρογνώμονες. Ήταν να γίνει συζήτηση. Δεν έχω ετοιμάσει κάτι ως και ο έχω όμως κάποιες ερωτήσεις. Εγώ είμαι τυχερή αλλά και άτυχη ενδεχομένως ε, για την Κομισιόν διότι ασχολούμαι, είμαι και μέλος της Επιτροπής ε, Δημοσιονομικού Ελέγχου. Οπότε το βλέπω από δύο προοπτικές, και από την πλευρά της απασχόλησης το θέμα και από την πλευρά του Δημοσιονομικού Ελέγχου. Ήμουν μάλιστα πρόεδρος μιας αποστολής της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου στην Ιταλία και επιλέξαμε δύο περιφέρειες, δύο περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα με, με υψηλά ποσοστά ανεργίας, Σικελία και Καλάβρια. Ε, και συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με αυτά που είπατε προηγουμένως για το ποιε αλλαγές πρέπει να λάβουν χώρα και πού πρέπει να βελτιωθούμε. Σίγουρα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην δημιουργία δυνατοτήτων σε διοικητικό επίπεδο, ε, την ενσωμάτωση κυρίω των συστημάτων πληροφορικης διότι αυτά που είδαμε εκεί ε, δεν ήταν και τόσο ενθαρρυντικά σε ό,τι αφορά τα συστήματα πληροφορική. Επίσης ενθαρρύνουμε τις περιφέρειες να συνδυάσουν την ε, ε, ε διάθεση των ε, κονδυλίων σε εθνικό επίπεδο με την συνδρομή, τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει εκεί να είμαστε πιο αποτελεσματικοί σε επίπεδο βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης χρειάζεται συνεργασία σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή η συνεργασία μπορεί να επαναφέρει την εμπιστοσύνη ε, στην αγορά εργασίας για τους νέους. Πρέπει να πω ότι ε, εμείς υπογραμμίζουμε ιδιαίτερα το, την ε, σημασία μιας προσέγγισης που να βασίζεται στην απόδοση, στην αποτελεσματικότητα αυτών των πρωτοβουλειών. Και έχω και κάποια ερωτήματα εδώ. Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα της πρωτοβουλίας απασχόλησης για τους νέους και της εγγύησης πώς μπορούμε να το μετρήσουμε, πώς μπορούμε να προσμετρήσουμε κατά πόσο τα χρήματα ε, πιάνουν τόπο. Μιλάμε για ε, τα διδάγματα, αλλά πώς, ε, πώς μετράμε αυτά τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ για την ΚΟΕ η κυρία Γκονζάλεθ Πένια, Πένιας. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Ναι, ακούστε να δείτε. Είναι σαφές νομίζω ότι η εγγύηση για τους νέους ήταν μια καλή πρωτοβουλία. Είναι μια καλή πρωτοβουλία, αλλά που δεν προγραμματίστηκε καλά. Μια απάντηση επίγουσα για ένα πρόβλημα το οποίο από ό,τι φαίνεται η Κομισιόν δεν το έχει αντιληφθεί στο σύνολό του. Όταν, όπως βλέπουμε, ε, όπως δείχνουν τα στοιχεία στην περιφέρεια της Ευρώπης, είναι δομικοί οι λόγοι της ε, ανεργίας των νέων, το παραγωγικό μοντέλο και αδυναμία του, ε, η μείωση της ζήτησης. Αυτό δεν μπορούμε να το ξεχνάμε. Βεβαίως η εγγύηση για τους νέους μπορεί ε, να κάνει κακό σε ό,τι αφορά την πολιτική απασχόληση των νέων, μεταξύ των οποίων και στα προγράμματα κατάρτισης. Θα ήταν κατάλληλο, θα ήταν πιο σωστό μάλλον να γίνει μια εφαρμογή λιγότερο βιαστική που να εγγυάται και την κάλυψη και τη χρηματοδότηση. Υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στο πρόγραμμα αυτό. Σε κάποιες χώρες είναι πολύ δύσκολη η εφαρμογή. Και μια πτυχή την οποία θα πρέπει να εξετάσει και το ελεκτικό συνέδριο στην επόμενη εκθεσή του για να μπορέσει αυτή η εγγύηση για τους νέους να είναι αποτελεσματική, θα πρέπει να βασιστεί στις βέλτιστες πρακτικές που θα έχουμε εντοπίσει. Ε, και εδώ θα ήθελα να στήσω τη γνώμη των εμπειρογνωμόνων. Ε, γιατί σε πολλές χώρες, όπως στη δική μου, στην Ισπανία, το πρόγραμμα βασίστηκε στις άμεσες ενισχύσεις των επιχειρήσεων. Αυτό ήταν καλό για τις επιχειρήσεις, αλλά όχι απαραίτητα για την πρόσληψη των νέων ανθρώπων που είναι στην ανεργία. Ή συχνά αφορά δραστηριότητε που ήταν ήδη προγραμματισμένε, οπότε δεν φέρνει κάτι καινοτόμο. Θεωρείτε ότι αυτά πρέπει να αποκλειστούν ω εναλλακτικέ. Ε, μήπως πρέπει να χρηματοδοτούνται μόνο προγράμματα τα οποία έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά του και την προσθετικότητά του και φέρνουν αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τους πράσινους η κυρία Χένκε. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για αυτήν την έκθεση. Τώρα είναι κάπως υπερβολικό να μιλάτε για καθαρή, για ξαφή μείωση της ανεργίας των νέων. Έχουμε κάποιες θετικές τάσεις, αλλά ας μην πέσουμε στην παγίδα τώρα της αυταρέσκειας, διότι εντάξει έχουμε απλά μια μικρή μείωση, είναι μια καλή αρχή. Έχω και εγώ κάποιες ερωτήσεις για τους πυρογνώμονες. Ε, κάποιοι συνάδελφοι ήδη αναφέρθηκαν. Το πρώτο που θέλω να ρωτήσω είναι, λέτε ότι 70% των νέων στους οποίους ε, ε, δίνεται μια προσφορά, υπάρχει μια προσφορά θέσης απασχόλησης, ε, η, έρευνα όμως αναφέρει, μετράει πόσο βιώσιμες είναι αυτές οι προσφορές. Είναι συμβόλαια για δύο-τρεις μήνες και μετά, ξανα, ε, και μετά επιστρέφουν στην ανεργία. Ε, αυτές οι θέσεις απασχόλησης είναι ε, είναι αξιοπρεπής, είναι επισφαλής, ε, είναι καλές συνθήκες εργασίας. Επίσης ε, υπάρχει το θέμα των της από χώρα σε χώρα, διότι πρέπει να δούμε τα αποτελέσματα που διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Υπάρχει το παράδειγμα της Ισπανίας, αλλά θα ήταν καλό να μας πείτε κι εσείς πού μπορεί κανείς να εντοπίσει βέλτιστες πρακτικές. Το όριο ηλικίας είναι 25 αυτή τη στιγμή. Ε, μήπως πρέπει να το ξαναδούμε αυτό, μήπως θα μπορούσαμε να το επεκτείνουμε στα 29, 30, διότι σε πολλά κρατημέλη ε, κάποιοι ακόμα σπουδάζουν μέχρι και τα 29, 30, είναι, αυτό συμβαίνει συχνά στη Γερμανία παραδείγματος χάρη. Και τέλος, ε, μίλησατε για τη μαθητεία και την ποιότητα ε, αυτών των προγραμμάτων μαθητείας. Θέλω να ρωτήσω, ε, δεν είναι τόσο μεγάλος ο αριθμός, 12,1% των προσφορών. Ε, θα προτείνατε ενδεχομένως οι μαθητίες και τα στάζ να, τα, να αφαιρεθούν για να μην υπάρχει αυτή η δυνατότητα αυτοί οι νέοι να πηγαίνουν τελικά από στάζ σε στάζ χωρίς τελικά να τους προσφέρει κάποιος μια βιώσιμη θέση απασχόλησης. Ευχαριστώ. Η κυρία Μελά και ο κύριος Μαχτά, ενδεχομένω δύο λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είναι σημαντικό ε, να δούμε λίγο πώς έχουν τα πράγματα. Τον Οκτώβριο του 2016 4.169.000 νέοι ήταν άνεργοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 18,4% εκ των οποίων 2.930.000 εντός της Ευρωζώνης. Και αυτό δείχνει ότι τα τρία τέταρτα των νέων άνεργων προέρχονται από την Ευρωζώνη. Το 2012 υπήρχαν εννέα ε, χώρες όπου η ενεργεία των νέων ήταν πάνω από 25%. Εξακολουθούν να είναι πέντε χώρες σήμερα όπου το ποσοστό ανεργίας των νέων είναι πάνω από 25% και χαίρουν ε, της ενίσχυσης των σχετικών προγραμμάτων. Το 2015 11 χωρίς 25% στην, στο Βέλγιο 22%, στην ε, Ισπανία 48%, στην Φιλανδία 22%, στη Γερμανία 24,6%, στην Ελλάδα 49,8%, στην Ιρλανδία 20,8% στην Ιταλία 40-33, στην πολωνια 20,75, στην πορτογαλια 31,95, στη Σλοβακία 26, στη Σουηδία 20,32. Μόνο η Γερμανία έχει ποσοστό ενεργείας των νέων κάτω από 10%. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2012 προσπαθεί να φρενάρει, να μετριάσει τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης που μαστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σπαταλά δισεκατομμύρια ε, προς τις χώρες ε, που έχουν πληγεί από αυτήν την μαζική ενεργεία των νέων. Τα σημαντικά ποσοστά ανεργίας των νέων σε 11 κράτη-μέλη αποδεικνύουν τα όρια σε επίπεδο αποτελεσμάτων των ε, συστημάτων αυτών, των προγραμμάτων αυτών, ιδιαίτερα στη Γαλλία. Σήμερα θέλει να ενισχύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα σύστημα το οποίο δεν έφερε πραγματικά αποτελέσματα και ούτε πρόκειται να φέρει στο μέλλον. Συμπερασματικά, Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ίσως τελικά να είναι ε, ο Δήμιος που αφού έχει θανατώσει το θύμα του, του βάζει επίδεσμους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει η κυρία Σαρτιέ. Ε, τέσσερα ερωτήματα έχω να θέσω προς τους πυρογνώμονες. Το πρώτο στις πηγές σας από τη Eurostat φαίνεται ότι αυτοί οι οποίοι εγκαταλείπουν το σχολείο ε, πρώιμα είναι λιγότερο το 2015 σχέση το 2008. Θα ήθελα να ξέρω όμως εάν αυτό το συνδέεται με την οικονομική κρίση. Δηλαδή είναι πιο δύσκολο να βρει κάποιος μια θέση εργασίας, να βρει θέση στην αγορά εργασίας και ίσως γι' αυτό οι μαθητές εγκαταλείπουν τα σχολεία νωρίτερα δεν εγκαταλείπουν τα σχόλια μάλλον νωρίτερα. Ε, θα πρέπει πριν να επιχαίρουμε να δούμε ποιες είναι οι αιτίες. Επίσης ε, βλέπουμε ότι από 16, μιλάμε για 16 εκατομμύρια τα οποία συμμετέχουν ε, στην εγγύηση για τους νέους, 10 εκατομμύρια όχι θέσεις απασχόλησης, έτσι. Μπορεί να είναι μαθητεία, μπορεί να είναι κατάρτιση, μπορεί να είναι στάζ. Συμφωνώ λοιπόν με τον Τέρι θα το παρακολουθήσουμε αυτό, τι θα γίνει μετά από δύο, τρία, τέσσερα χρόνια, διότι εκεί θα φανεί, ε, θα φανούν τα συμπεράσματα. Το τρίτο τώρα, είπατε ότι ήταν σημαντικές οι συμπράξεις μεταξύ διαφορών υπηρεσιών στα πλαίσια αυτής της εγγύησης για τους νέους. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό μάλλον ήταν ε, υπηρεσίες ε, ε, που δεν ήταν πραγματικά, πραγματικά αποτέλεσμα συμπράξεων. Και επίσης υπήρξε ένα πρόβλημα αναγνωσιμότητας μεταξύ της εγγύησης για τους νέους, της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων. Ε, πώς θα το διορθώσουμε αυτό. Ε, εδώ συμφωνώ με τη Μαρτίνα Διαμπάλοβα προηγουμένως. Πρέπει να δείξουμε την αποτελεσματικότητα της πολιτικής μας, ναι, να τη δείξουμε, αλλά πρέπει επίσης να είναι αναγνώσιμο αυτό. Ευχαριστώ. Θα δώσω και πάλι το λόγο για Σόστροβα και στη συνέχεια θα τροποποιήσω κάπως τη σειρά που είχε προβλεφθεί έτσι ώστε οι δύο εμπειρογνώμονε να μπορέσουν να παρέμβουν και αυτό θα μας επιτρέψει στη συνέχεια να έχουμε ακόμα λίγο χρόνο και να έχουν και αυτοί χρόνο βεβαίως να απαντήσουν στα ερωτήματα που τέθηκαν. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Βολό. στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων. Τα επόμενα θέματα, εκεί θέλω, το επόμενο θέμα, εκεί θέλω το λόγο. Καλώς λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Άνια Μέγικορτ, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα μιλήσω για την ε, πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Ξέρετε ότι είχα εγώ την ευθύνη της αξιολόγησης των πρώτων αποτελεσμάτων πέρσι για την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά και την Αγγλία ειδικότερα, αλλά έχω και άλλα αξιολογήσεις προγραμμάτων για την νεολαία αναλάβει. Σύντομα, ο σχεδιασμός της πρωτοβουλίας έχει καλυφθεί λίγο πολύ, πολύ σύντομα θα σας τον υπενθυμίσω. Κύρια ευρήματα της υλοποίησης, μάλλον αυτό που σας ενδιαφέρει περισσότερο θα είναι τα αποτελέσματα και τα επιτεύγματα, οι ε, αδυναμίες, ε, τα πλεονεκτήματα και συμπεράσματα με συστάσεις. Πώς ε, έχει σχεδιαστεί λοιπόν η πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ακούσαμε εν συντομία το πώς έχει σχεδιαστεί. Σε περιφερειακό επίπεδο ορίστηκε η αιρεσιμότητα, επίπεδο ΝΑΤΣ 2, 20 κρατημέλη, χρηματοδότηση, με βάση τα δεδομένα της ανεργίας των νέων του 2012. 25% των ανέργων, των νέων ήταν άνεργοι, ή χωρίς ε, δραστηριότητα που μάλιστα έχει φτάσει στο 30%. Βλέπετε τα κράτη που δεν είχαν ε, επιλεξιμότητα και για την πρωτοβουλία αλλά και για την εγγύηση. Η πρωτοβουλία για την απασχόληση χρηματοδοτεί μέτρα που αφορούν τους νέους νίτς, αυτούς δηλαδή που δεν είναι ούτε στο εκπαιδευτικό σύστημα της απασχόληση, ούτε σε μαθητεία ή πρακτική εκπαίδευση μέχρι τα 25 ή τα 29 όπως επέλεξαν ορισμένα κράτη-μέλη ετηλικίας που έχουν κατοικία σε, σε επιλέξιμη περιοχή. Σημαντικό είναι να γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει χρηματοδότηση για προληπτικές δράσεις, πριν να καταστεί δηλαδή ένας νέος που βρίσκεται σε τέτοιο κίνδυνο, νέος της κατηγορίας NEET. όπως ξέρετε έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα ε, του Κοινωνικού Ταμείου 2014-2020 και τα λειτουργικά προγράμματα που διαχειρίζονται οι ε, αρχές διαχείρισης. 6,4 δις η χρηματοδότηση, συνολικά 3,2 ειδικά για την πρωτοβουλία και 3,2 από τις εθνικές ε, πιστώσεις για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Στη χρηματοδότηση 1,1 κράτη-μέλη για το κομμάτι του κοινωνικού ταμείου. Αποδέκτες. Η Ισπανία, ένα τρίτο της χρηματοδότησης, η Ιταλία, η Γαλλία, η Πολωνία και μετά σε μικρότερα ποσά η Σλοβενία, η Κύπρος και η Τσεχική Δημοκρατία. Και θα δείτε με βάση τους ειδικούς κανόνες για την ταχεία υλοποίηση, αποδέσμευση των κονδυλίων, ε, διευκόλυνση χρηματοδότηση κτλ. Δεν φαίνεται να είχαν ιδιαίτερη απόδοση γιατί οι λόγοι στην καθυστέρηση της υλοποίηση δεν ήταν τόσο οικονομική όσο διοικητική σε επίπεδο επιλέξιμων κρατών μελών. Τι ξέρουμε λοιπόν για την υλοποίηση της πρωτοβουλία. Τι κάνουν τα κράτη με τα χρήματα αυτά. Η έρευνά μας ε, έλαβε χώρα τον Νοέμβριο του 2015, έχει περάσει αρκετός καιρός, αλλά δεν νομίζω ότι θα έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικά ως προς τις δραστηριότητες των κρατών μελών. Ε, προτείνουν λοιπόν υποστήριξη με τρία ή περισσότερα μέτρα για την ε, εγγύηση απασχόλησης. Επιτοπλίστων στοχεύουν στην απόκτηση επαγγελματικής πείρας ή μαθητείας, 83% των διαχειριστικών αρχών έχουν πρώτη επαγγελματική εμπειρία επιλέξει, 72% μαθητεία πρακτική εξάσκηση, 65% ε, ποιοτικά μαθήματα και επίσης ενίσχυση νέων επιχειρηματικών ε, σε ποσοστό κοντά στο 55%. Και... Κάποιες χώρες κάνουν κάπως ε, διαφορετικά πράγματα, νομίζω η Ιταλία και η Γαλλία που έχουν μια εθνική ε, πολιτική θητεία θα λέγαμε με χρηματοδότηση και επίσης γύρω στο 60-70% της χρηματοδότησης στη Γαλλία πηγαίνει σε συμβουλευτικές υπηρεσίε αναζήτησης εργασίας. Επίσης δεν υπάρχει μέτρο για να αποτρέψει τους νέους από το να πέσουν σε αυτή την κατάσταση και ένα άλλο πράγμα το οποίο πρέπει να ξέρετε είναι ότι όλες οι χώρες δήλωσαν ότι έχουν εξατομικευμένα σχέδια δράσης, μία από τις πρότασεις ε, που σχετίζονται με την χρηματοδότηση αυτή, αλλά βεβαίω το τι εννοεί κάθε χώρα διαφέρει. Κάποιε χώρε μιλάνε για πακέτα μέτρων, τρία διαφορετικά μέτρα, στα οποία έχουν πρόσβαση οι νέοι. Άλλε χώρε έχουν αξιολόγηση των αναγκών και σχετικέ δραστηριότητε. Ε, τέθη πριν ένα ερώτημα για την καινοτομία. Κοιτάμε την καινοτομία των ε, μέτρων σε διάφορα κράτη-μέλη και είδαμε ότι ενώ υπάρχουν κάποια παραδείγματα καινοτομία, ε, και κάποιων οργανισμών που είναι καινούργοι και δεν έχουν πρόσβαση στο χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, βλέπουμε πως ένα μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης του προγράμματος αυτού της εγγύησης για την Ελλάδα ε, πηγαίνει σε υφιστάμενα μέτρα τα οποία ενισχύονται. Π.χ. στην Ιρλανδία έχουμε ενίσχυση των μέτρων που υπήρχαν στο παρελθόν, στη Γαλλία ενισχύονται υφιστάμενα μέτρα, σε πολλά κράτη-μέλη. Και ένας παράγων είναι ο χρόνος. Η στιγμή δηλαδή μεγάλοι οργανισμοί με εμπειρία μπόρεσαν να κάνουν προσφορές για αυτά τα κονδύλια και οι μικρότεροι οργανισμοί, ίσως πιο καινοτόμοι, χρειάζονταν περισσότερο χρόνο και βρέθηκαν σε μειονεκτική θέση. Οπότε, τι ξέρουμε για τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής, ε, πόσοι νέοι δηλαδή έχουν εμπλακεί μέχρι στιγμής και ποια είναι τα αποτελέσματα και πόσοι έχουν ενταχθεί στην εκπαίδευση ή απασχόληση. Λοιπόν, 2014 είχαμε μια πάρα πολύ αρχική υιοθέτηση και δεν είχαμε δεδομένα. Μετά το 2015 έχουμε δεδομένα από τις εκθέσεις εφαρμογής και γνωρίζουμε ότι γύρω στους 500.000 συμμετέχοντες ε, συμμετείχαν ε, τότε. Το 2016 δεν έχουμε αξιόπιστα δεδομένα. Προφανώς υπάρχει η δημοσίευση της Κομισιόν η οποία συνοψίζει τα αποτελέσματα του εγγύηση τη συνολία που λέει πω 1,4 ε, εκατομμύρια νέοι έχουν εμπλακεί, αλλά εγώ θα έλεγα ότι είναι μάλλον χαμηλότερο το νούμερο. Π.χ. για του λόγου ε, που ανέφερε η Ισπανίδα βουλευτής ότι μεγάλος αριθμός νέων στην Ιταλία και η Ισπανία είναι εγγεγραμμένοι αλλά δεν ωφελούνται από το πρόγραμμα. Παραδείγματο χάρη στην Ιταλία το Μάρτιο του 2016 έχουμε 640.000 νέους που είχαν εγγραφεί αλλά μόνο 220.000 ε, παρεμβάσεις έλαβαν χώρα, οπότε το 1 τρίτο, δεν μιλάμε για άτομα, παρεμβάσεις. Ε, μπορεί να είναι άτομα δηλαδή τα οποία έχουν λάβει περισσότερες παρεμβάσεις και να είναι ακόμη λιγότεροι οι νέοι που έχουν καλυφθεί από το πρόγραμμα και θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες τον Μάιο-Ιούνιο με την νέα ετήσια έκθεση εφαρμογής που θα υποβάλουν τα κράτη-μέλη. Υπήρχαν κάποιες αρχικές ε, πρωτοβουλίες στην εμπλοκή ευπαθών ομάδων, οι εθνικές αξιολογήσεις ε, που ξεκίνησαν στο τέλος 2015 που λέγαν πως υπήρχαν κάποιες δυσκολίες παρόμοιες με την εγγύηση για τους νέους και η έρευνα την οποία κάναμε στο τέλος του 2015 έλεγε ότι αρχικά τα κράτη-μέλη ασχοληθήκαμε με τους πιο νέους 15 με 24 ετών άνδρες ε, 51% και με όσους είχαν τουλάχιστον δεύτερο βάθμα εκπαίδευση και βεβαίως αυτοί οι οποίοι ήταν ανενεργοί και δεν είχαν ίσως εγγραφεί στα ταμεία ενεργείας. Αυτό το οποίο είναι ενδιαφέρον επίσης είναι η κάλυψη κάτι το οποίο προέκυψε νωρίτερα νομίζω ε, προφανώς ε, δεν μπορούμε να καλύψουμε όλους τους νέους οι οποίοι θα είναι επιλέξιμοι σε όλα τα κράτη-μέλη, είναι σε περιφερειακή βάση, αλλά είναι ενδιαφέρον να συγκρίνουμε το ποσοστό των ατόμων που έχουν εμπλακεί στο πρόγραμμα μέχρι στιγμή. Ε, Ιούλιο 2016 έχουμε τα πιο πρόσφατα δεδομένα και το ποσοστό των ατόμων στις χώρες Λοιπόν, αν δείτε εδώ πέρα τον πίνακα, βλέπουμε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλε διαφορέ μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τα ποσοστά ατόμων που δεν εκπαιδεύονται ή δεν δουλεύουν και έχουν εμπλακεί στο πρόγραμμα αυτό. Βλέπουμε Λετωνία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Γαλλία, ένα στου πέντε νεαρού, στου νεαρού που δεν ε, εκπαιδεύονται ή εργάζονται στην πρωτοβουλία αυτή, ενώ Ρουμανία και Ηνωμένο Βασίλειο δεν είχαν ξεκινήσει, αλλά και μικρότερα ποσοστά σε Σλοβακία, Τσεχία κτλ. Έχω εξαιρέσει την Ιταλία και την Ισπανία γιατί δεν γνωρίζουμε πόσοι νέοι συμμετείχαν, όπως σας είπα και πριν. Αποτελέσματα λοιπόν, αποτελέσματα μέχρι το τέλος του 2015 για να σας δώσω μια ιδέα για τα ποσοστά των ατόμων που συμπλήρωσαν ε, το πρόγραμμα ή όσους ε, ε, κάνουν μια μετάβαση. Λοιπόν, το τέλος του 2015 γύρω στους 500.000 άτομα είχαν λάβει μέρος σε προγράμματα σε μέτρα του προγράμματος, γύρω 40% ε, είχαν ολοκληρώσει με εκείνη τη στιγμή. Αυτό δεν σημαίνει ότι μόνο 40% ε, θα το ολοκληρώσουν, απλά ακόμη πολλοί ήταν σε, στο πρόγραμμα το οποίο ήταν εν εξελίξη. Και βεβαίως ε, σκοπεύουμε κατά μέσο όρο να έχουμε 70% ποσοστό ολοκλήρωση. Λοιπόν, από αυτούς οι οποίοι συμπλήρωσαν το πρόγραμμα, 80.250 έλαβαν μια πρόσφορα είτε εκπαίδευση είτε εργασίας και 109.000 άτομα βρήκαν ε, εκπαίδευση ή εργασία. Και αυτό μάλλον οφείλεται στο ότι κάποιοι βρίσκουν μόνοι τους ε, δουλειά ή εκπαίδευση ή ε, ότι μπορεί να εκμεταλλευτούν κάποια άλλη ευκαιρία από μόνοι τους και το ποσοστό αυτό μετάβασης δεν είναι τόσο κακό γιατί τα περισσότερα κράτη-μέλη στοχεύουν να κάπου μεταξύ 25 και 50% να έχουν προσφορές εκπαίδευση εργασία. Και βεβαίω σε το ζήτημα τη ποιότητα των προσφορών και όλοι αναρωτιόμαστε και δεν ξέρουμε. Και αυτό γιατί πολλά κράτη-μέλη καθορίζουν διαφορετικά την ποιότητα των προσφορών. Κοιτάμε την δικιά μας μελέτη, είδαμε πώς θα καθορίζουν τα κράτη-μέλη και κάποια κράτη-μέλη λένε ότι είναι μια βιώσιμη προσφορά, άλλοι λένε ικανοποιητική προσφορά, αλλά δεν ξέρουμε στην πραγματικότητα κατά πόσον είναι. Υπάρχει μια ένδειξη της διάρκειας, το οποίο μας δίνει ε, βεβαίως μια έννοια του μακροπρόθεσμου αποτελέσματος έξι μήνες μετά το λήξη του προγράμματος. Αυτό θα φανεί βεβαίως στην αιτήσια έκθεση ένα συγκεκριμένο παράδειγμα από την ε, Σλοβενία που μου ζητήθηκε να συγκρίνω με την Ισπανία γιατί η Σλοβενία συχνά θεωρείται ως κάτι το θετικό στην ε, ανεργία των νέων. Λοιπόν, η πρωτοβουλία αυτή. Ένα λόγο για τον οποίο ήταν επιλέξιμη η Σλοβενία με μια συνολική αξία του προγράμματο γύρω στα 20 εκατομμύρια ευρώ είναι η μικρότερη κατανομή από όλα τα επιλέξιμα κράτη-μέλη και παραδείγματο χάρη 100 εκατομμύρια εξοδεύει η ίδια η χώρα σε ένα έτος οπότε μιλάμε για μικρό σχετικά ποσό και χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά για την πρωτοβουλία, η πρώτη πρόκληση όπως λέγεται, ένα πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης για άτομα τα οποία μπαίνουν πρώτη φορά στην αγορά εργασίας και στόχο είχε 3.000 ε, νεαρούς και βλέπουμε ότι στο τέλος Ιουνίου 2016 είχε φτάσει σε 2.000 ε, νεαρούς ε, και βεβαίω ε, αρκετοί από αυτούς είχαν βρει κάποια πρόσβαση. τέσσερα άτομα, Βεβαίω, αυτό μάλλον είναι, οφείλεται στο ότι πολλοί ήταν ακόμα μέσα στο πρόγραμμα, στην παρέμβαση και θα βελτιωθούν τα αποτελέσματα αργότερα. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην Σλοβενία υπάρχει πολύ στοχευμένη επιρροή του προγράμματος ε, της ε, πρωτοβουλίας αυτής, δηλαδή ο αριθμός των ατόμων είναι οριακό σε σχέση με τις ανάγκες που υπάρχουν, δηλαδή γύρω 40.000 άτομα στην ομάδα αυτή την ηλικιακή στην χώρα. Λοιπόν, ποια είναι τα ισχυρά και τα δύναμα σημεία της πρωτοβουλίας. Ε, βασικό ισχυρό σημείο είναι ότι έχει διαθέσει επιπρόσθετη χρηματοδότηση για μέτρα απασχοληση των νέων, ειδικά σε κάποια που διαφορετικά δεν θα υπήρχε χρηματοδότηση, είτε γιατί δεν είναι πολιτική προτεραιότητα. Οπότε, δεύτερο βασικό σημείο, έχει πολύ θετικό αντίκτυπο σε όλα τα κράτη-μέλη. Επίση, η χρηματοδότηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μια κάποια ευελιξία, αν και συχνά σα λένε ότι δεν έχουν έτσι τα πράγματα οι διαχειριστικέ αρχέ, αλλά θεωρητικά μπορεί να προσαρμοστεί στις τοπικές και περιφερειακές ανάγκες και γενικά υπάρχει μια θετική αντιμετώπιση. Προφανώς ε, υποστηρίζει την εισαγωγή της εγγύησης για τους νέους σε κάποιες χώρες και ε, μπορούμε να συζητήσουμε την άλλη επικάλυψη στις ερωτήσεις και βέβαια διευκολύνει τη μετάβαση από πολιτικές αγοράς εργασίας οι οποίες βασίζονταν κυρίως ε, στην προσφορά σε μια πολιτική που ενισχύει την ζήτηση. Ποιες είναι οι αδυναμίες τώρα του προγράμματος. Όπως είπαμε, ο χρόνος, το πολύ μικρό χρονικό διάστημα για την εφαρμογή, ε, πρόκειται για μια ατυχή στιγμή γιατί οι διαχειριστικές αρχές προετοιμάζονταν για την επόμενη περίοδο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και ήταν δύσκολο να εντάξουν κάπου αυτή την πρωτοβουλία. Πρόκειται λοιπόν για ένα μέσο χρηματοδότησης δεν είναι ένα μέτρο, εξαρτάται από τα μέτρα που παρέχονται στα κράτη-μέλη. Και υπάρχουν βεβαίως κάποια ζητήματα που δείχνει η εθνική αξιολόγηση σε κάποια κράτη-μέλη και μετά υπάρχει η δυσκολία του να ταυτοποιηθούν οι νέοι οι οποίοι αποκλείονται. Επίσης ε, θεωρείται γραφειοκρατική η πρωτοβουλία ακόμα και σε σύγκριση με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο γιατί απαιτούνται επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία και γίνεται αγώνας πραγματικά παραδείγματος χάρη ε, για κάποιους νέους ε, να αποδείξουν τον τόπο που είναι προαπαιτούμενο και επίσης ε, είχε βασιστεί σε ποσοστά ανεργίας του 2012 και σε κάποιες περιφέρειες η κατάσταση έχει αλλάξει. Είναι λιγότερη ας πούμε ναι. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν στο μέλλον. Μπορούμε να το δούμε αυτό σε ερωτήσεις γιατί τελειώνει και ο χρόνος. Αλλά προφανώς συζητήσαμε ήδη την παράταση της ε, περίοδου εφαρμογής πέρα από το 2018 και με περισσότερη χρηματοδότηση. Νομίζω είναι σημαντικό αυτό, αλλά σημαντικό επίσης είναι να δούμε ποια θα είναι η εφαρμογή. Δεν νομίζω ότι τα κράτη-μέλη ωφελούνται συνολικά με τα περισσότερα κονδύλια. Πρέπει να αξιολογηθεί ποιε περιφέρειες αυτή τη στιγμή χρειάζονται περισσότερα κονδύλια και για ποιου είδου δραστηριότητε. Διαφορετικές έρευνες πρέπει να γίνουν και μια παρόμοια τέτοια κονδύλια στο μέλλον, πρέπει να δούμε να, πώς θα αυξηθεί η αποτελεσματικότητα μέσω καλύτερης συμβατότητας με το χρονοδιάγραμμα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και φυστάμενε δραστηριότητες. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε για αυτές τις πληροφορίες, για αυτή τη σημαντική δουλειά αξιολόγησης που έλαβε χώρα. Το είδαμε και στην παρουσίασή σας, έχουμε πολλά στοιχεία περιφερειακά. Θα περάσουμε τώρα μια άλλη πτυχή σε σχέση με την ανάλυση που έχει να κάνει με τις ιδιαιτερότητες της περιφερειακής, τα στοιχεία δηλαδή που έχουν να κάνουν με την περιφερειακή κάλυψη και πιο συγκεκριμένα την κατάσταση στην Ισπανία. Η Ελβίρα Γκονσάλεθ Γκάγκο θα κάνει τη σχετική παρουσίαση. 15 λεπτά παρακαλώ. Thank you. Thank you very much for me to here. Ευχαριστώ που θα μας με καλέσατε να παρουσιάσω αυτή την περίπτωση της Ισπανίας που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα με πολλές διαφορές σε σχέση με αυτά που έχουν εξηγηθεί εδώ. Εγώ είμαι εδώ ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πραγματογνωμοσύνης. Εργαζόμαστε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεθνής Απασχόλησης, για ζητήματα αγοράς εργασίας και έχουμε κάνει μια σειρά από έρευνες που σχετίζονται με ε, την νεολαία Σε τέσσερα μέρη χωρίζεται η παρουσίασή μου. Θα εξηγήσω λίγο τις, ε, τους διακανονισμούς εφαρμογής της ε, πρωτοβουλίας για, τους, ε, για την απασχόληση των νέων. Των Γέι το ονομάζουμε εμείς, έτσι θα το ονομάζω από εδώ και πέρα. Να σας εξηγήσω λοιπόν πώς εφαρμόζουμε την ΓΕΙ και την εγγύηση για τους νέους. Στη συνέχεια θα κάνω κάποια σχόλια για την εφαρμογή της ΓΕΙ μετά θα σας μιλήσω για τις εξελίξεις την εξέλιξη μάλλον της ανεργίας μεταξύ των νέων και τέλος θα αναφερθώ σε κάποια σημαντικά ευρήματα και συστάσεις. Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της ΓΕΙ ξεκινήσαμε τον Απρίλιο του 2013 στα πλαίσια της ε, στρατηγικής για την επιχειρηματικότητα και την ε, ε, απασχόληση των νέων για, τα, για τους νέους 130 ετών. Δεν περιζόμαστε δηλαδή στους νέους κάτω των 24. Το Δεκέμβριο του 2013 η κυβέρνηση υπέβαλε ένα σχέδιο για την εγγύηση των νέων, για την εφαρμογή τη εγγύηση για του νέου, που είναι μια αντιγραφή τη στρατηγική για την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση των νέων που έχει ξεκινήσει το ίδιο έτο νωρίτερα τον Απρίλιο. Τον Δεκέμβριο του 2014, ένα χρόνο αργότερα, το επιχειρησιακό πρόγραμμα για την απασχόληση των νέων εγκρίθηκε και αυτό το επιχειρησιακό πρόγραμμα έχει αφιερωθεί αποκλειστικά στην εφαρμογή της εγγύησης για τους νέους και η ΓΕΗ, η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων, ε, περιλαμβάνεται σε αυτό το επιχειρησιακό πρόγραμμα. Η... Ε, το, 80% του, της χρηματοδότησης για την εγγύηση των νέων αφορά την, απασ... την, την πρωτοβουλία απασχόλησης των νέων. 2,7 δισεκατομμύρια δηλαδή στην χώρα μας 943 εκατομμύρια είναι το ΓΕΙ ε, στην χώρα μας, το μεγαλύτερο ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε χρηματοδότηση του τάξη των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Κάποια σχόλια τώρα για τους δικαιούχους της πρωτοβουλίας αυτής, της εγγύης για τους νέους και της ΓΕΙ. Εμείς αποφασίσαμε αρχικά ότι η ομάδα ε, στην οποία αφορά το σύστημα είναι ηλικίας 16 έως 24, όμως τον Ιούλιο του 2015 το επεκτείναμε έως τα 29 έτη εφόσον ξεπερνάει το 20% το ποσοστό ανεργίας. Οι απαιτήσει επιλεξιμότητας, τα κριτήρια επιλεξιμότητας που αναφέρονται ε, αρχικά ήταν τόσο αυστηρά περιόρισαν σε μεγάλο βαθμό την συμμετοχή των νέων. Τον Δεκέμβριο του 2016 λοιπόν επανεξετάσαμε τις προϋποθέσεις αυτές, τις καταστήσαμε πιο ευέλικτες, ιδιαίτερα ε, η προϋπόθεση ότι αυτοί που είναι εγγεγραμμένοι ε, στην υπηρεσία για τη δημόσια απασχόληση ε, μπορούσαν να εγγραφούν πιο εύκολα στο πρόγραμμα. Όλες οι ισπανικές περιφέρειες είναι επιλέξιμες για την ΓΕΗ, ενώ αρχικά είχαν, το είχαμε αφιερώσει, οι, μισοί πόροι μάλλον έχουν, αφιερωθεί στις περιφέρειες. Ξέρετε ότι περιφέρειες ε, στη χώρα μας έχουν πολλές αρμοδιότητες με μια αποκεντρωμένη διοίκηση έτσι οι μισοί πόροι έχουν αφιερωθεί στις περιφέρειες αυτές με βάση βεβαίως τις ανάγκες τους. Η υπόλοιπο στασμός γίνεται κεντρικά, ενώ τα σημεία κλειδιά για την Ισπανία είναι ότι έχουμε μια πολύ καλή έχουμε δημιουργήσει μια πολύ καλή σύμπραξη με μια σειρά από ευλεγόμενε φορεί. Έχουμε ένα ευρύ δίκτυο σημείων ενημέρωσης, το, Εθνικό Ινστιτούτο Νεολαίας, ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ε, η YMCA, το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης που ασχολείται με το συντονισμό ε, με τις τοπικές διοικήσεις το Δεκέμβριο του 2016 και αυτό είναι σημαντικό το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Υγείας Κοινωνικών Υπηρεσιών και Ισότητας συμμετέχουν και αυτά σε αυτήν την σύμπραξη. Το Υπουργείο Παιδείας έως τώρα, ναι, μάλλον αρχικά δεν συμμετείχε. Ήταν το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών που συμμετείχε. Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η Ισπανία έχει προβεί και μεταρρυθμίσει να εφαρμόσει την ΓΕΗ ευθυγραμμιζόμενη ε, στις διάφορες μορφές ενεργούς πολιτικής στην εργασία για να βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ της κεντρικής ε, διοίκησης και των περιφερειών. Σε ό,τι αφορά τώρα την εφαρμογή της ΓΕΗ, όπως ανέφεραν οι προηγούμενοι μιλητές, η εφαρμογή είναι πίσω σε σχέση με το μεσόρο της Ένωσης και σε ό,τι αφορά την κάλυψη και σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση έχω πάντως την εντύπωση ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος το 2016. Παρ' όλα αυτά το ποσοστό κάλυψης για ε, την και ομάδα 15 με 29 αυτή τη στιγμή το Φεβρουάριο του 2017 ήταν της τάξης του 32% περίπου. Βεβαίως δεν έχουμε επίσημα στοιχεία μετά το, το τέλος του 2015. Βασιζόμαστε λοιπόν στα δεδομένα για, που αφορούν όλους τους νέους που έχουν εγγραφεί στο σύστημα, στο σύστημα και αξιολογούμε ε, αυτήν ακριβώς την ηλικιακή ομάδα. Είμαστε πολύ πίσω σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήταν 37% ε, αλλά έχουμε διπλασιασμό σε σχέση με το Φεβρουάριο του 2016. Έχω λοιπόν την εντύπωση ότι η φάση εφαρμογής έχει προχωρήσει, ιδιαίτερα το 2016 με γοργά βήματα, άλλα αποτελέσματα τώρα από τη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Έχουμε επίση πολύ μεγάλε ανισότητε, πολύ μεγάλε αποκλήσει από περιφέρεια σε περιφέρεια. Στην Ανδαλουσία, στην Ναβάρα, στην Καλήθεια, στι Αστούρια έχουμε πάνω από 40%, ενώ σε άλλε περιφέρειε όπω η Μελίγια και η Θέουτα είμαστε κάτω από το 20% σε ό,τι αφορά την κάλυψη. Είμαστε κοντά στο 75% ε, σε ό,τι αφορά ε, τα θετικά αποτελέσματα, πολύ μεγαλύτερη, μεγαλύτερο από το μέσο όρο τον ευρωπαϊκό, διότι μόνο 40% ε, των προσφορών έχουν να κάνουν με την απασχόληση, οι υπόλοιπε προσφορές έχουν να κάνουν με δεύτερη ευκαιρία εκπαίδευσης, ε, κατάρτισης, Τώρα σε ό,τι αφορά την βιωσιμότητα της ένταξης, εδώ είναι πάλι ο δείκτης αντίστοιχος με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής, 37% στην Ισπανία, 40% στο σύνολο της Ένωσης. Λοιπόν, γιατί υπάρχει καθυστέρηση και γιατί είναι περιορισμένη εφαρμογή. Υπήρξε μια σύγχυση αρχικά και μια βεβαιότητα σε ό,τι αφορά το οποίο μπορεί να είναι επιλέξιμος για τη γέη και για την εγγύηση των νέων και επίσης υπήρχε μια επικάλυψη στις διάφορες προγραμματικές περιόδου καθώς και καθυστερήσεις της έγκρισης των προγραμμάτων. Το Μάιο του 2016 είχαμε την έγκριση, αυτό σημαίνει ότι πολλά από τα ενδιάμεσα όργανα ήδη εφάρμοζαν μέτρα χωρίς να γνωρίζουν αν τα μέτρα αυτά θα είναι επιλέξιμα τελικά. Ένας δεύτερος λόγος είναι η ευρύτερη οικονομική συγκυρία, έχουμε την εξυγέννηση δημοσιονομική. Από το 2007 έως το 2013 ο προϋπολογισμός για την πολιτική απασχόληση μειώθηκε κατά 30% και μιλάμε για μια εποχή σημαντικής αύξησης της ανεργίας. Οπότε οι πολιτικές ε, για την απασχόληση μειώθηκαν κατά 68% ανά άτομο. 10% ανά άτομο ε, σε σχέση με το ποσοστό που διατίθεται στη Δανία και 30% σε σχέση με το ποσοστό ε, που διατίθεται στη Γαλλία και κάτι παρεμφερές στη Γερμανία. Αυτό σημαίνει ότι η ΓΕΙ δεν μπόρεσε να αναπληρώσει αυτήν την πολύ σημαντική μείωση των δημοσιονομικών πόρων. Ένας άλλος λόγος για τη μειωμένη, την, την μη πρόοδο, εν περιπτώσει, είναι η έλλειψη διοικητικών δυνατοτήτων που οι δημόσιες αρχές ε, παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στη σύμπραξη αυτή και είναι υπεύθυνε για την εφαρμογή της ΓΕΗ. Έλλειψη καινοτομία επίσης έχει υποθεί και στο παρελθόν. Επικεντρώθηκαν αποκλειστικά οι δραστηριότητε οι δράσεις στην πλευρά της προσφοράς. Μόλις 30% των προσφορών έχουν να κάνουν με κάτι ε, άλλο από αυτό, οπότε ουσιαστικά αυξάνεται ο ανταγωνισμό για τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας, ε, και συχνά οδηγούμαστε στι θέσει εργασία με χαμηλότερου μισθού και πιο ε, επισφαλεί συνθήκε εργασία αναφερθώ τώρα στην εξέλιξη της ανεργίας και της απασχόλησης ε, των νέων στην Ισπανία. Εδώ αριστερά στο γράφημα βλέπετε την εξέλιξη της ανεργίας των νέων στην Ισπανία σε απόλυτους αριθμούς. Θα το διαβάσω εγώ για σας. Το βασικό μήνυμα είναι ότι η ανεργία των νέων αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο ανθρώπους από το 2008 έως το 2010 η μισή από αυτούς τους νέους ανθρώπους είχαν χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Κατά την ανάκαμψη, από το 2013 δηλαδή και μετά έως το 2015, περίπου περίπου έχουμε περίπου 400 λέει μιλήτρια λιγότερους άνεργους βλέπουμε όμως ότι περίπου 2 εκατομμύρια νέοι άνεργοι είχαν χάσει τη δουλειά τους στην πρώτη φάση της κρίσης από το 2008 στο 2010. Όμως, από το 2013 έως το 2016 μόλις 21.000 θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν για τους νέους. Με πολύ μεγάλες αποκλήσεις από περιφέρεια σε περιφέρεια, η Καστία, Ελαιών ε, έχουμε 40% ε, μείωση της ανεργίας των νέων, όμως στη Βαλένθια μόλις 6% κτλ. λοιπά. Η ποιότητα τώρα έγινε σχετική αναφορά για την ποιότητα των θέσεων απασχόλησης. Οι λίγοι νέοι άνεργοι που βρήκαν δουλειά ε, βρήκαν θέσεις απασχόλησης με πολύ ε, χειρότερες συνθήκε εργασία, ε, ε, προσωρινά συμβόλαια, χαμηλή μισθή. ...25% μείωση των μισθών για τους νέους. Οι βασικές προκλήσεις τώρα για την Ισπανία. Η Ισπανία θα πρέπει να αυξήσει, να βελτιώσει την εφαρμογή της ΓΕΙ... ...και αυτό πρέπει να γίνει με ένα ολοκληρωμένο σύστημα πληροφοριών δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί το σύστημα αυτό και είναι απαραίτητο να ολοκληρωθεί για να υπάρξει μια σωστή παρακολούθηση, να υπάρχει διαφάνεια, να υπάρχει αξιολόγηση. Πρέπει να ε, βελτιωθεί επίση ο συντονισμό μεταξύ όλων των ενδιάμεσων ε, φορέων που συμμετέχουν στην, στην, ε, στο σύστημα, να ενισχυθεί η εφαρμογή στι περιφέρειες που έχουν μείνει πίσω, πρέπει να αυξηθούν οι δυνατότητες οι διοικητικές με, ποσοστό, με, με προσωπικό καλύτερα καταρτισμένο, να έχουμε μια εφαρμογή περισσότερων μέτρων που έχουν να κάνουν με τη ζήτηση και εδώ υπάρχει μεγάλη διαφορά με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν επενδύουμε επαρκώς ε, σε μέτρα που έχουν να κάνουν με τη ζήτηση. Μια άλλη πρόκληση είναι να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες των νέων που ε, διατρέχουν τον κίνδυνο της φτώχειας ή και του κοινωνικού αποκλεισμού. Σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να ε, παραταθεί παρά η περίοδος ε, εφαρμογής για την απορρόφηση των κονδυλίων. Δεν θα προλάβει να απορροφήσει όλα τα κονδύλια η Ισπανία έγκαιρα και θα πρέπει να μείνει η χρηματοδότηση στο ίδιο επίπεδο του 2018, λαμβάνοντα υπόψη ότι η ΓΕΙ αποτελεί 80% της χρηματοδότησης ε, του προπολογισμού της εγγύησης για τους νέους. Έως το 2018, οπότε θα μένει 20% μέχρι το 2023, θα έχουμε σημαντική μείωση λοιπόν. Αυτά είμαι στη διαθεσία για να απαντήσω στα ερωτήματά σας. Donc on vient de voir des éléments Ευχαριστώ πολύ. Είδαμε λοιπόν τα στοιχεία αξιολόγησης και μια συγκεκριμένη εικόνα της κατάστασης στην Ισπανία θα λάβουν οι εισηγητές και οι εισηγητής και σκιώδης ε, το λόγο. Πάνω λεπτό καθένας. Παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την παρουσίαση. Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία που μας παρουσιάσατε. Και αφού άκουσα την ε, παρουσίασή σας, πιστεύω ότι θα πρέπει να ομολογήσουμε πως είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα τα σχετικά με την επιτυχία του προγράμματος. Ασφαλώς, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, επενδύθηκαν ε, σημαντικά ποσά για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και βλέπουμε ότι τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικά επίπεδα απορρόφησης. Δεν μπορούμε όμως να κατηγορούμε για τα πάντα τις ε, ευρωπαϊκές υπηρεσίες. Θα πρέπει να διερωτηθούμε πόσο συγκεκριμένη ήταν η περιγραφή από πλευρά των κρατών μελών των ίδιων, γιατί εκείνα καλούνται να υλοποιήσουν στις χώρες τους τα προγράμματα. Εάν λοιπόν να συζητήσουμε την συνέχιση ή τη διακοπή των προγραμμάτων αυτών ή την αναστολή τους και νομίζω ότι όλοι θα θέλαμε να προχωρήσουμε σε κάτι περισσότερο μάλλον, θα πρέπει να πούμε ναι. Το πρόγραμμα έχει φέρει θετικά αποτελέσματα, έχει φέρει πολλά καλά. Αλλά φαντάζομαι ότι με τις ε, διαπιστώσεις σας μπορούμε και στο μέλλον να έχουμε και περισσότερες διασμεύσεις και περισσότερη διαφάνεια για τη χρήση των κονδυλίων και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Για τα ποσά λοιπόν, έστω να προβλέπονται σημαντικά ποσά. Αλλά πρέπει να ξέρουμε τι είδου λύσει είναι αυτέ, βραχυπρόθεσμε ή μακροπρόθεσμε. Γιατί δεν μπορούμε να δημιουργούμε θέσει εργασία με χρηματοδότηση. Πρέπει πάνω απ' όλα να μεριμνήσουμε για την αποκατάσταση τη οικονομία. Για να δώσουμε καλέ και μόνιμε λύσει. Και θέλω ιδιαίτερα να τονίσω κάτι πολύ σημαντικό. Ότι όταν έχει ολοκληρωθεί ένα πρόγραμμα για τους νέους, θα πρέπει να υπάρχει επαρκή κάλυψη των θέσεων εργασία στην αγορά. Όχι να του αφήνουμε ξεκρέμα. Στου ε, σοσιαλιστέ δημοκράτε δεν έχουν κανέναν. Ε, η CM επίση. Κυρία Λαμπάιωα, καλύτερα. Ναι, πρόεδρε, ευχαριστώ. Και πολύ σύντομα, κάτι που ανέφερα και νωρίτερα, για την ε, μέτρηση της αποτελεσματικότητας πρέπει οπωσδήποτε να κοιτάξουμε την στόχευση σε μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Και θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας. Εσείς που έχετε δει στην πράξη πώς υλοποιούν τα κράτη-μέλη, μακροπρόθεσμα τα αποτελέσματα αυτά πώς μπορούμε να τα προσμετρήσουμε, γιατί βραχυπρόθεσμα μόνο βλέπουμε την εικόνα. Η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων επίσης, το λέτε κι εσείς. Θεωρείτε ότι έχει μεγάλο ποσοστό γραφειοκρατικής επιβάρυνσης. Τι βήματα λοιπόν θα μπορούσαν να ληφθούν για να διευκολυνθεί ο δικαιούχος όταν θέλει να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση. Και επίσης δεν πρέπει να στοχεύουμε στις εταιρικέ σχέσεις μόνο για την απασχόληση, την εκπαίδευση κλπ. Όλες οι πολιτικές που αφορούν την νεολαία θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους για να έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Και επίσης, η υποστήριξη που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κράτη και περιφέρειες έχει τεράστια σημασία πέραν των εθνικών ή περιφερειακών προσπαθειών. Ιδιαίτερη σημασία έχει η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μπορεί έτσι να κλείσει και το κενό στην υλοποίηση αλλά και να βελτιώσει την αποδοτικότητα. Άλλο τόσο άλλως όμως έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει προσφέρει σημαντική αρρωγή στα κράτη και στις περιφέρειες. Ο Πρόεδρος ευχαριστώ. Χένκε. Ε, ευχαριστώ και εγώ τους ομιλητές. Πρέπει να παραδεχτώ ότι ειδικά το παράδειγμα της Ισπανίας ε, μου έδειξε πως αυτό το οποίο πρέπει να δούμε είναι η συνοχή της πολιτικής. Γιατί αφενός, αν έχουμε μείωση των πολιτικών ε, της αγοράς εργασίας κατά 68% που δεν είναι ε, αποκλειστικά, αλλά οφείλεται και στο ότι η Ισπανία ήταν στο πρόγραμμα και έχουμε εξυγίανση του προπολογισμού που κόβει κονδύλια και από την άλλη ε, ερχόμαστε με κοινοτική χρηματοδότηση που είναι σημαντική και χρήσιμη, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορεί να αντισταθμίσει πλήρως το κενό που δημιούργησε μια άλλη ευρωπαϊκή πολιτική. Νομίζω ότι γινόμαστε ασυνάρτητοι και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορέσει να λύσει η πρωτοβουλία αυτή. Και πρέπει να το πάρουμε σοβαρά. Και ακριβώς θα πρέπει να δούμε πώς θα λύσουμε το πρόβλημα της ενεργείας των νέων, ειδικά στις χώρες του Νότου. Πρέπει να δημιουργήσουμε δουλειές χωρίς επενδύσεις ε, στην οικονομία και ποιοτικέ θέσει εργασία ε, δεν θα μπορέσουν οι νέοι να μπουν στην αγορά εργασίας, αν ε, δεν υπάρχουν δουλειέ. Ε, νομίζω αυτό προέκυψε και όταν μιλούσατε για τα αποτελέσματα στην Ισπανία. Έχω και μία ερώτηση και για τους δυο σας. Σε σχέση με τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Είπατε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερες έρευνες. Ήδη είχα την εντύπωση ότι από τα ευρήματα που έχετε ε, δεν έχω μια γενική εικόνα γιατί υπάρχουν τόσες πολλές αναπάντητες ερωτήσεις και ήθελα να σας ρωτήσω πότε θεωρείτε ότι θα έχουμε μια πληρέστερη εικόνα και τι έρευνα θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει για να αξιολογήσουμε όχι μόνο την εφαρμογή της ε, πρωτοβουλίας αυτής συνολικά, αλλά συγκεκριμένα να δούμε τις βέλτιστες πρακτικές. Γιατί νομίζω ότι στο παράδειγμα της Ισπανίας βλέπουμε ποιες είναι από τις προκλήσεις, αλλά μπορούμε να δούμε και άλλα παραδείγματα όπου τα πράγματα πήγαν καλά και να μάθουν και άλλα κράτη-μέλη κάτι. Σας ευχαριστώ. Να υπάρχει κάποιος από το ΙΕΝΕΦ, η κυρία Σωτονβέ, για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, λέει κυρία Σόντροβα. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια και μια ερώτηση. Νομίζω ότι οι πρωτοβουλίε αυτέ, η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων και η εγγύηση για του νέου, ε, σωστά στοχεύουν στου νέου ε, άνεργου ε, που δεν εκπαιδεύονται. Με το παράδειγμα της Ισπανίας βλέπουμε ότι είναι σωστή η αισθίαση των πρωτοβουλίων αυτών και δεν πρέπει να υποτιμάμε ότι είναι πολύ σημαντικά αυτά τα προγράμματα, αλλά νομίζω ότι είναι και κατακαιρματισμένες αυτές οι πρωτοβουλίες. Κοιτώντας ε, ας πούμε, το δίκτυ προστασίας των νέων μεταξύ 17 και 30 ετών. Έχουμε τις δύο πρωτοβουλίες, ε, το Σώμα Αλληλεγγύης, ε, Τέσσερα προγράμματα δηλαδή που δρούν παράλληλα και η νέα αυτή πρωτοβουλία που προετοιμάζεται. Λοιπόν, πρέπει νομίζω να δούμε την ε, αποτελεσματικότητα όλου αυτού του συστήματος. Όπως σας είπα, σωστή η προτεραιότητα, αλλά κατακαιρματισμένη. Αυτές είναι οι πρωτοβουλίες που βασίζονται σε προτάσεις της Κομισιόν. Το Κοινοβούλιο στηρίζει τον γενικό στόχο, δηλαδή τα κράτη-μέλη να παρέχουν καλύτερη εκπαίδευση και εμπειρία στην εργασία και αναζήτηση εργασίας. Αλλά τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε θα πρέπει να συντονίζονται καλύτερα ακόμα και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό το οποίο θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι η δική σας η άποψη για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης που επίσης προετοιμάζεται και η ανακοίνωση της Κομισιόν λέει ξεκάθαρα ότι η πρωτοβουλία για τους νέους και η εγγύηση για τους νέους θα είναι τα δύο προγράμματα τα οποία κυρίως ε, θα δημιουργήσουν αυτό το νέο μέσο. Νομίζω ότι έχετε ενημερωθεί γι' αυτό και το δεύτερο ερώτημα, με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αναφέρατε ότι στην Σλοβενία γίνεται ένα έργο στα 20 εκατομμύρια ευρώ. 2.000 ε, άτομα λαμβάνουν μέρος με 10.000 ευρώ ανά άτομο, πολύ γενναιόδωρο. Μπορείτε να μου πείτε, θεωρείτε ότι ε, αρκεί αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. 10 λεπτά μας μένουν περίπου. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Βερνέ γιατί τέθηκαν μια σειρά από ερωτήσεις. Βεβαίως όλες οι ερωτήσεις που τέθηκαν δεν μπορούν να απαντηθούν σε 10 λεπτά. Παρ' όλα αυτά κάντε μια προσπάθεια απαντήσετε σε κάποιες ερωτήσεις και δώσετε και την δυνατότητα ε, στους εμπειρογνώμονε να μιλήσουν και αυτοί για ένα-δύο λεπτά ο καθένας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κάπω ε, δύσκολη θέση για να επιλέξω μεταξύ των ερωτήσεων γιατί αυτά τα οποία αφορούν ε, την ε, πρωτοβουλία για την απασχόληση μπορώ να τα απαντήσει συνάδελφο. Εγώ θα ασχοληθώ με το θέμα τη εγγύηση για του. νέου. Πρώτα απ' όλα έγινε μια παρατήρηση για το ότι τα δεδομένα της εφαρμογής ε, ήταν κάπως ασυνεπή, ειδικά το ποσοστό κάλυψης και οι επιτυχημένες ε, έξοδοι. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι καθώς η εγγύηση για την νεολαία είναι μια νέα πολιτική, σχετικά η συλλογή των δεδομένων ε, επίσης είναι στην αρχή. Οπότε έχουμε αυτή τη στιγμή δεδομένα μόνο από το 2014 και 2015 Κάτι το οποίο σημαίνει ότι χρειαζόμαστε λίγο χρόνο για να είναι αξιόπιστα τα δεδομένα, αλλά του λεχθέντος γεγονός είναι ότι η πρόοδος είναι άνηση, αυτό είναι ήδη φανερό, αλλά αυτό οφείλεται επίσης στο ότι και η κατάσταση διαφέρει πολύ από χώρα σε χώρα. Για το συγκεκριμένο ερώτημα που αφορά το ποσοστό κάλυψης και εξόδου, βλέπουμε ότι κάποια κράτη-μέλη επέλεξαν να καλύψουν περισσότερους νέους, αλλά μετά βεβαίως η αποτελεσματικότητα της εγγύησης των νέων ε, όσον αφορά το ποσοστό επιτυχίας δεν είναι τόσο μεγάλη. Άλλα κράτη-μέλη πρώτα προσέφεραν μια εγγύηση σε μικρό ποσοστό των ατόμων αυτών, αλλά μετά είναι σε θέση να έχουν υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο παρατηρούμε στη συλλογή των δεδομένων. Έγινε ένα σχόλιο για συγκεκριμένα προγράμματα για την εγγύηση για την νεολαία, ότι δεν είναι αποτελεσματική, καινοτόμο και πρέπει να βοηθούν αυτά τα πράγματα. Ε, Εστιάζοντα δηλαδή στην πλευρά τη πολιτική, ε, είμαστε συνεχώ σε επαφή με τα κράτη-μέλη και όχι μόνο μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και του ΕΜΚΟ του υψηλότερου επίπεδου, αλλά έχουμε και επαφές σε επίπεδο εργασίας, έχουμε το δίκτυο των συντονιστών και μάλιστα το λέμε στα κράτη-μέλη όταν βλέπουμε ότι κάποια προγράμματα πρέπει έτσι, κάπως να βελτιωθούν. Ε, το τελευταίο Ε, θα πω ότι η Κομισιόν μπορεί να καταργήσει πλήρως προγράμματα, αλλά μπορεί να συμβουλεύσει κάποια κρατημέλη να βελτιώσουν τα προγράμματα. Μετά. μια ερώτηση για το πώς μετράμε την ε, βιωσιμότητα των προσφορών και ειδικά των προσφορών εργασίας που είναι πιο δημοφιλής έχουμε κάποια δεδομένα παρακολούθησης, οπότε συλλέγοντας δεδομένα υπάρχουν, συλλέγονται δεδομένα για το τι συμβαίνει στα άτομα που εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία 6, 12 και 18 μήνες μετά από την αποδοχή της προσφοράς. Ε, το πρόβλημα είναι ότι επειδή είμαστε στην αρχή της εφαρμογής έχουμε δεδομένα μόνο για τους 6 μήνες. Αλλά όσο περνάει ο χρόνος θα έχουμε περισσότερα δεδομένα. Και έτσι θα μπορέσουμε να δούμε σε ποιο βαθμό τα πρόγραμματα αυτά είναι βιώσιμα. Το εάν τώρα οι προσφορές για εργασία υπάρχουν καλές συνθήκες εργασίας, είναι πολύ σημαντική ερώτηση και οφείλω να πω ότι δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό τόνισα ότι είναι πολύ σημαντικό να συζητήσουμε περαιτέρω με τα κράτη-μέλη το θέμα της ποιότητας πώς θα διασφαλίσουμε την ποιότητα των προσφορών και αυτή τη στιγμή η Κομισιόν συνεργάζεται με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας για να καθορίσουμε την ποιότητα των προσφορών αλλά και να δούμε την δυνατότητα του να συζητήσουμε ε, τις προδιαγραφές ποιότητας ε, με τα κράτη-μέλη στην ΕΜΚΟ την Επιτροπή Αποσχόλησης αλλά το αποτέλεσμα εξαρτάται από τα κράτη-μέλη. για την ερώτηση για τις βέλτιστες πρακτικές. Δεν ξέρω πόση ώρα έχω. Α, τελείωσε ο χρόνος. Τότε σύντομα το θέμα του ορίου ηλικία. Αυτό το αποφασίζουν τα κράτη-μέλη και τα μισά κράτη-μέλη μάλιστα αποφάσισαν να το ανεβάσουν στα 29. Να προσφέρουν εγγύηση για την νεολαία μέχρι τα 29. Ε, τέλος, αν δεν θέλει να παρέμβει σε αυτό η Κομισιόν. Και τέλος υπόθηκε ότι αν θα πρέπει να αφαιρέσουμε τις μαθητείες γιατί αποτελούν μόνο το 12% γεγονός είναι ότι σε πολλά κράτη-μέλη μαθητεία θεωρείται δουλειά και την καταγράφουν ως δουλειά οπότε ε, υπάρχουν ε, και μαθητείες εκεί πέρα αλλά εν πάση περιπτώσει η Κομισιόν δεν σκοπεύει να αφαιρέσει τις ε, μαθητείες από την εγγύηση για την δουλειά. Θα δώσω τώρα τον λόγο συνάδελφο. Thank you. This on. Yes. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να καλύψω 5 λεπτά σε 1,5, 5 ε, λεπτό. Όπως και για τις εγγυήσεις των νέων υπάρχει ένα μεσοπρόθεσμο αποτέλεσμα, ένας δείξης μεσοπρόθεσμα αποτέλεσματος για ε, περίπου 6 μήνες μετά. Πολλά από τα κράτη-μέλη που γνωρίζουν κάνουν προσπάθειες έτσι ώστε να κάνουν καλύτερε εκτιμήσεις του αντικτύπου τη παρέμβαση, κάνουν αξιολογήσεις και αυτό θα είναι σημαντικό στο μέλλον. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμω ότι σε πολλά κράτη-μέλη η κατάσταση για τα δεδομένα δεν είναι καλή για αυτές τις αξιολογήσεις και κανείς ε, δεν πρέπει να υποχρεούται να το εφαρμόσει. Καλό είναι πάντως να έχουμε όσο γίνει περισσότερες πληροφορίες και αποτελέσματα. Δεύτερον, τι πρέπει να αλλάξει για να είναι λιγότερο διοικητικά επαχθές. Υπάρχουν δύο επίπεδα. Το πρώτο είναι αυτό που είπα στα συμπεράσματά μου εάν υπήρχε καλύτερη ευθογράμμιση με, το ESF, διότι οι, αρχές διαχείρισης αλλά και πολλές οργανώσεις, οι οργανώσεις μάλλον ε, που εμπλέκονται φέρνουν αποτελέσματα, τότε θα είχαμε ένα λιγότερο διοικητικά επαχθές πρόγραμμα. Επίσης για να καταστεί σαφέστερο πώς τα κριτήρια, πώς η πλησιμότητα των νέων μπορεί να αποδειχθεί. Το ξέρουμε αυτό και από την Ισπανία και από την Αγγλία όμως. Πολλοί από τους παρόχους θεωρούν ότι πρέπει να δώσουν στοιχεία για τη διαμονή, ε, αλλά υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία και είναι ευθύνη της Κομισιόν ή και της Αρχής Διαχείρισης να είναι σαφέστερη ότι μπορούν να ζητηθούν αποδεικτικά στοιχεία λιγότερο αυστηρά. Πότε θα έχουμε μια σαφέστερη εικόνα. Το Μάιο-Ιούνιο θα έχουμε τα στοιχεία του 2016 ε, για την ε, πρωτοβουλία απασχόληση των νέων. Δεν ξέρω πότε θα τα λάβετε εσεί, αλλά η Κομισιόν θα τα έχει σίγουρα τότε και τότε θα έχουμε και την ε, επισκόπηση 2015-2016 και επίσης υπάρχει θεματοβέλη των πρακτικών. Η αξιολόγηση ε, οι θα την έχουμε στο τέλος του 2018 δυστυχώς, όταν τελειώσει το πρόγραμμα. Ε, θα δώσουν πληροφορίες βέβαια τότε για βέλτιστες πρακτικές αυτές οι αξιολογήσεις, αλλά κάποιες πληροφορίες αυτές μπορούν, μπορεί ενδεχομένω να τις έχουμε νωρίτερα και βέβαια είναι σημαντικές πληροφορίες. Ε, δεν έχω πολλές πληροφορίες για ε, την, ε, την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Ε, δεν ξέρω πώς μπορεί να συμπεριληφθεί, με το, να, να συνδυαστεί με το European Solidarity Fund Funds, το δική μας πρωτοβουλία, έπρεπε να έχουν ήδη διατεθεί τα χρήματα, οπότε δεν βλέπω πώς μπορεί να υπάρξει εδώ συνδυασμό, να μπορεί να πει η Κομισιόν κάτι περισσότερο και τέλος, το πόσα χρήματα διατέθονται, για τους νέους ε, ανα κεφάλι, ανα άνθρωπο. Αυτό εξαρτάται. Για κάποιους νέους που είναι μακριά, πολύ μακριά από την αγορά εργασίας, θα πρέπει κανείς να επενδύσει περισσότερα χρήματα από 1000 ευρώ ας πούμε. Εξαρτάται ε, τι θέλουμε να πετύχουμε με το μέτρο και ποια, ποια είναι η ομάδα στόχος. Για τα άτομα παραδείγματος χάρη με αναπηρίες προφανώς ε, κοστίζει κάτι περισσότερο. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά έχουν μείνει. Σχόλια που αφορούν τη συνοχή στην, ε, στον περιορισμό των αποκλήσεων. Έχουμε 68% σε συνδυασμό της χρηματοδότησης των δύο μέσων και έχετε δίκιο. Βλέπαμε ότι δεν προχωρούσε από την εποχή εκείνη η υπόθεση. Και αυτό δείχνει, ε, εξηγεί και γιατί ήταν τόσο αργή η κίνηση. Ε, σχόλιο ότι δεν μπορούμε να δημιουργούμε θέσεις εργασίας. Μα είναι τεράστιες οι ανάγκες σε ε, εκπαίδευση και δεν έχει κανένα νόημα να προβλέπουμε το ένα πρόγραμμα μαθητείας μετά το άλλο όταν δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας γιατί μόνο δυσφορία προξενεί. Αυτό που προβλέπετε τώρα στην Ισπανία είναι κίνητρα για προσλήψεις. Χαμηλότερη συμμετοχή του εργοδότη στην κοινωνική πρόνοια, αλλά και άλλα συστήματα για συμμετοχή στο χώρο εργασίας, στην αγορά εργασίας των νέων. Παραγωγικό όμως ε, δεν αποδειχθεί κανένα από αυτά. Πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο και αν να, κάνουμε, να φτιάξουμε τις εργασίες, πρέπει να είναι καλές αυτές. Οι επιδοτήσεις μάλλον αποτελούν απλώς έναν τρόπο μεταφοράς κονδυλίων προς επιχειρήσεις. Στην ε, περιφερειακή διάσταση τώρα νομίζω ότι για την Ισπανία ειδικά μπορούμε να στηριχθούμε στην περιφερειακή διάστηση, Έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Ιδιαίτερα στην Καταλωνία, με ανθρώπους δραστήριους, νέους, που δουλεύουν καλά και με τις αρχές τις τοπικές, φέρνουν αποτέλεσμα. Και αυτό μπορεί να βελτιώσει και την αποτελεσματικότητα και θα έλεγα και τη διαφάνεια βέβαια. Πρέπει να ενισχυθεί η διαφάνεια. Δεν είναι καθόλου γνωστή η εγγύηση για την απασχόληση των νέων στην ε, ε, Ισπανία. Σε σχέση δε με αυτήν δεν έχω ιδέα αν υπάρχει κάποιο συσχετισμός με το Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Δουλέψαμε πάρα πολύ καλά. Κάναμε πολλαπλές και πολλοί επίπεδες αναλύσεις. Αποδείχθηκε πόσο κρίσιμα είναι αυτά τα θέματα και οι στόχοι που εξυπηρετούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σας ευχαριστώ όλους και ιδιαίτερα το τμήμα θεματικών μελετών που θα ετοιμάσει και το σχετικό, τη σχετική τεκμηρίωση. Ευχαριστώ τους ομιλητές μας εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης Έμπλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τους ειδικούς, ζητώντας πάντα συγγνώμη για τον λίγο χρόνο που είχαμε στη θέσή μας. Πάντα είναι ο χρόνος λιγοστός. Ευχαριστώ τους συναδέλφους, βουλευτές και δι αυτούς που έμειναν μέχρι τέλους. Ευχαριστούμε και τους διερμηνείς, λέει ο Πρόεδρος και οι ευχαριστώ. σας ευχαριστούν. 3 Απριλίου έκτακτη συνεδρίαση στο Στρασβούργο, 11 και 12, εδώ στις Βρυξέλλες. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλό βράδυ.